Uh, Καλησπέρα σε όλους. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Να σας πω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα της ε, συνεδριασής μας διότι μαζί μας βρίσκονται μέλη της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης του ΠΟΕ και είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια κοινή, μεκτή συνεδρίαση. Καλωσορίζω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας και όπως ίσως τα γνωρίζετε ήδη, έχει υποθεί αρκετές φορές, η ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου είναι αυτό που μας συνδέει με την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ Και η προσπάθεια αυτή για τη διακοινοβουλευτική συνέλευση ξεκίνησε το 2002. Είναι ένα μεγάλο κοινό εγχείρημα. Υπάρχουν 22 μέλη. Οι περισσότεροι βρίσκονται εδώ, στην αίθουσα, στο πίσω μέρος. Να σας καλωσορίσω θερμά στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αύριο θα έχετε τη δική σας την σύνοδο και όπως είχε γίνει και πέρσι αποφασίστηκε ακριβώς να οργανωθεί συνάντηση της ομάδας της Steering Committee εδώ στις Βρυξέλλες, όπως είχε γίνει και πέρσι. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ΠΟΕ, τον ομόλογό μας στην Διευθυντική Επιτροπή και μέλος της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΠΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για το θερμό σας καλωσόρισμα. Ε, ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στο κοινοβούλιο από το οποίο έφυγα πριν από 14 περίπου χρόνια. Ήμουν εδώ κάποια δεκαετία περίπου. Επειδή όμως ε, ο Όλιβερ Ντόνελ που είναι ο αρμόδιος για τα θέματα αυτά, αρμόδιος από τον Καναδά, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε που μας προσκαλέσατε στην, ε, στην συνεδρίαση αυτή και του συναδέλφου σα που μα δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε. Σωστά το περιγράψατε. Εδώ έχουμε συνάντηση τη Διευθυντική ε, Επιτροπή, τη κοινοβουλευτική συνέλευση. Και συζητούμε κυρίω εμπορικά θέματα, τα οποία είναι τόσο επίκαιρα αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να προσπαθήσει να μεταστρέψει την κοινή γνώμη και να ακουστεί η φωνή μας ώστε να επηρεάσουμε πολλά από τα σημαντικά ζητήματα που εξελίσσονται και βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζεται και θα διαδραματίσετε στι εμπορικέ διαπραγματεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ μέρου των συναδέλφων μου, στο πίσω μέρο τη αίθουσα και του κυρίου Σέργεϊ Τσέρνακοφ που μας παρακολουθεί. Πραγματικά έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψει και ελπίζω ότι και αύριο θα έχουμε συμμετοχή και από εσάς με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και αύριο και στην τέταρτη συνδιάσκεψη, τη διυπουργική. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Συμπροεδρεύουμε σε αυτή την ε, συνάντηση. Τώρα το θέμα αυτού του τμήματος της συνεδριασής μας αφορά κάτι που ήδη σας ανακοίνωσα ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις των ΠΟΕ. Για να μας μιλήσει, έχουμε μαζί μας έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο, τον κύριο Ρούφους Γέρτσα, που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τον προσκαλέσαμε να μας ενημερώσει για τις πρόσφατες εξελίξεις στο επίπεδο του ΠΟΕ. Κύριε Γέρτσα, είστε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από το 2002 οι τομεί αρμοδιότητά σα αφορούν την επίλυση διαφορών, την ε, πρόσβαση στη βιομηχανική αγορά, την πνευματική διοκτησία, τι ε, προσχωρήσει και τι διευκολύνσει του εμπορίου. Επίση, είστε επιφορτισμένο με καθήκοντα εσωτερική διοργάνωση και εποπτεία του ΠΟΕ και του προπολογισμού 230 εκατομμυρίων δολαρίων του ΠΟΕ. Ε, Επίση, είσαστε υπεύθυνο για τη συνεργασία με τον Αμερικανό πρέσβη τη Συμφωνία Γκάτ και συμμετέχετε στι σχετικέ συζητήσει στην Ουάσιγκτον. Στο Μίνσκ πρόσφατα συμμετείχατε σε συζητήσεις στη Βουλή Και βεβαίω στην Ουάσιγκτον είσαστε επιφορτισμένου με την υποεπιτροπή εμπορίου τη κυβέρνηση εκεί. Σα ευχαριστούμε και λοιπόν κύριε Γέρτσα που ήρθατε. Είμαστε Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε λοιπόν ε, εν ώψη της διευπουργικής ε, Συνδιάσκεψης του Δεκεμβρίου. Ε, μετά από την σημερινή μας τη σημερινή σας παρέμβαση. Θα, το, δώσω το λόγο σε μέλη όχι μόνο στα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά και στα μέλη της Διευθυντικής Επιτροπής. Παρακαλώ να συμμετάσχετε στην όλη συζήτηση, γιατί είναι πολύ καυτό το θέμα του ΠΟΕ. Κύριε Γέρτσα, και πάλι ευχαριστώ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Μορέιρα. Ευχαριστώ και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και τα μέλη της IPU. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Η συνάντηση αυτή πραγματικά σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην πορεία των σχέσεων του ΠΟΕ με τους βουλευτές. Μια σχέση που διαρκώς προχωρά και εξελίσσεται και ενδυναμώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Έχουμε κάνει πολλά από την πρώτη μας συνάντηση στο Σιάτλ το 1999. Εκεί συμμετείχατε ενεργά και μια δεκαετία αργότερα οι σχέσεις του ΠΟΕ με τους βουλευτές έχουν ε, πραγματικά εξελιχθεί. Συναντιόμαστε συστηματικά σε επίπεδο IPU με τους βουλευτές για να ανταλλάσσουμε απόψεις και πληροφορίες για τα ωφέλη του ανοίγματο των αγορών και των ε, μεγαλύτερων ευκαιριών θέλουμε να προσφέρουμε ε, με εμπορικούς κανόνες και εμπορικές οργανώσεις για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ε, αλληλεπίδραση του ΠΟΕ με την κοινοβουλευτική δράση η κοινοβουλευτική διάσκεψη, συνέλευση μάλλον του ΠΟΕ είναι για μας πολύ σημαντική και από τη σκοπιά της δικής σας Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν καταρτήσει ένα πρόγραμμα δράσης, όπως ξέρατε είχαμε διπουργικέ συναντήσεις ήδη στο Κανκούν, τη Βρυσέλλες, το Χονγκ και στη Γενέβη και προσβλέπουμε στην ενεργό σας συμμετοχή στην διπουργική που θα γίνει αργότερα φέτος. Βεβαίως, οι βουλευτές διαδραματίζουν δικό ρόλο τα ξέρω, όπως είπατε κι εσείς, πολύ καλά αυτά, γιατί ήμουν μέρος του ε, προσωπικού, του συμβουλευτικού προσωπικού του Αμερικανικού Κογκρέσου για 9 χρόνια στην Washington. Ξέρω πώς επηρεάζουν οι ψηφοφόροι τις κυβερνητικές αποφάσεις, το κυβερνητικό σύστημα και καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να μεταφράζουμε σε εγχώρια εσωτερική πολιτική τις διεθνείς αποφάσεις και δεσμεύσεις. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορούμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας και στο μέλλον σε αυτήν την κοινή προσπάθεια όπως είπα, ως υπεύθυνη λήψης πολιτικών αποφάσεων σήμερα, δεν θα εκπλαγείτε αν ξεκινήσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες δυσκολίες ακόμα με την παγκόσμια οικονομία. Δεν έχουμε ξεφύγει από τις δυσκολίες, οι αριθμοί της ανάπτυξης είναι πολύ μικροί και τα ποσοστά ανεργίας πολύ ψηλά. Υπάρχουν σοβαρέ απειλέ σε τομεί όπω η επισητιστική ασφάλεια. Υπάρχει το ζήτημα του πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσει όπω οι κλιματικέ αλλαγέ και πολλά άλλα στοιχεία. Δυστυχώ δεν είναι πολλά ή πολύ καλά τα νέα ούτε στην εμπορική πλευρά του θέματος. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τους παγκόσμιους αριθμούς εμπορίου του ΠΟΕ για το 2012 και ετοιμάζουμε αυτούς το 2013 και είχαμε μια αύξηση μόνο του 2% το 2012. την ανάπτυξη που θα συνεχιστεί και το 2013. Εκεί προβλέπουμε 3,3 ανάπτυξη μόνον. Κάτω του 20 ετούς ε, συναθρισμένου στόχου του 5%. Υπάρχουν όμως κάποια καλά νέα, ιδίως στις χώρες μετάβασης και τις αναπτυσσόμενες. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές προβλέπεται να αναπτυχθούν να τριπλασιαστούν και να τετραπλασιαστούν ω προ την ταχύτητα σε σχέση με τι αναπτυγμένε χώρε. Το 2014 προβλέπουμε να αυξηθούν κατά 7,5%. Οι οικονομίε αυτέ δεν θα αναπτυχθούν μόνο οι ίδιε, αλλά θα ε, κινητοποιήσουν και την ε, παγκόσμια ανάκαμψη. Αλλάζουν λοιπόν ε, τα στοιχεία ε, στο παγκόσμιο σκηνικό, διότι πριν από 20 χρόνια 16% του διεθνού εμπορίου γινόταν στο βόρειο ημισφαίριο και το 30% ήταν το εμπόριο από το βορρά προ το νότο. 10% του παγκόσμιου εμπορίου ήταν ανάμεσα στι χώρε του νότου μεταξύ του. Μέχρι το 2020 περιμένουμε το εμπόριο στο νότο να φτάσει το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Βλέπετε πόσο εξελίσσονται τα πράγματα πώς ε, επηρεάζονται όλες οι χώρες, αλλά και πώς είναι διαφορετική η σύνθεση των ε, βιομηχανικών κλάδων παγκοσμίων πολλές και αλλαγές στις τεχνολογίες και τις μεταφορές που οδήγησαν στην ε, αύξηση των παγκόσμιων τιμών και αξιών και μέσω αυτής της αλλαγής οι αναπτυσσόμενες χώρες μπόρεσαν να δυσδύσουν καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία. Το εμπόριο δεν είναι πλέον κάτι που αφορά μόνο την πώληση τελικών προϊόντων υπηρεσιών σε άλλη χώρα, αλλά η ανταλλαγή τη δράση τη παραγωγή μεταξύ χωρών, παγκόσμιων προϊόντων πλέον. Μιλάμε για προστιθέμενη αξία με τη συμβολή όλων στα διάφορα στάδια τη παραγωγή ή με την παροχή υψηλή ποιότητα ε, υπηρεσιών. Μια άλλη θετική εξέλιξη στο επίπεδο του διεθνού ε, εμπορίου έχει να κάνει με το τι κάνουν οι κυβερνήσει ω τώρα, οι οποίες απήχαν από τον προστατευτισμό τον προστατευτισμό στο εμπόριο και τον έλεγχο των ε, οικονομικών δυσκολιών που αποπειρώνται από το 2008. Αυτά έχουν να κάνουν με τους κανόνες, της προδιαγραφές και το σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης του ΠΟΕ. Ελπίζουμε να, δια... να παραμείνουμε πιστοί στις υποσχέσεις μας προς τις αγορές. Βεβαίως ε, το ευάλωτο και το αβέβαιο της παγκόσμιας ανάκαμψης ε, ε, σχετίζεται και με τις σοβαρές απειλές που ελοχεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό που για μας είναι σαφές στον ΠΟΕ είναι ότι οι αγορές πρέπει να παραμείνουν σχετικά ανοιχτές. Χρειάζονται στρατηγικές από την κάθε χώρα για την προώθηση και την διατήρηση της ανάπτυξης μέσω μεγαλύτερης οικονομικής αλληλο... αλληλεξάρτησης και αλληλοσυσχετισμού. Πρέπει να παραμείνουμε σε ε, παγρύπνηση για να βεβαιωθούμε ότι οι οικονομικές ανάγκες λαμβάνονται υπόψη στον καταρτισμό πολιτικών. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γύρο της Ντόχα, όπως θα γνωρίζετε όλοι, το θέμα αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο παρά την τεχνοκρατική προσπάθεια να επιτύχουμε σύγκληση. Συνολικά η συμφωνία είναι κάτι το ανέφικτο. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι στον Παλί η διπουργική διάσκεψη ίσως είναι μια ε, ευκαιρία για να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη, τουλάχιστον σε τρία σημεία, εμπορικές διευκολύνσεις, γεωργία και αναπτυξιακά συμφωνίες μπορεί να έχουν και εμπορικό νόημα και να τονώσουν την ανάπτυξη, δίνοντας μια καλύτερη προοπτική, προοπτική μεγαλύτερης ανάπτυξης και αγοραστικής δύναμης για πολλές ε, ε χώρες. Για τις εμπορικές διευκολύνσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, τις καθυστερήσεις και τα απαγορευτικά γραφειοκρατικά όρια που αυτή τη στιγμή αποτελούν φραγμούς για το διεθνές εμπόριο. Ε, το κόστος της διακίνησης αγωθών ε, στον πλανήτη φτάνει 1,83 δολάρια ετησίως. Ένα δέκατο της αξίας του συνολικού όγκου εμπορευμάτων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αντιμετωπιστεί. Ε, το να μειωθεί το κόστος του εμπορίου θα αποδώσει ωφέλη σε όλους, διότι όσο λιγότερα δαπανώνται για να καλυφθεί το κόστος των συνελλαγών, τόσο περισσότερα θα εξοικονομούνται για να ωφελούνται οι καταναλωτές, η παραγωγή. Αυτό θα ωφελήσει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ε, χώρες που εξαρτώνται από την ε, εύκολη πρόσβαση στις αγορές, τις περίκλειστες χώρες. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις εμπορικές διευκολύνσεις είναι ότι υπάρχει σχέση της υλοποίησης από δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει αναπτυσσόμενες χώρες με την τεχνική στήριξη μπορεί να τους προσφερθεί για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και για να έχουν πραγματικά την ε, ικανότητα, την ευκαιρία να προβλέψουν τα μέτρα που θα επιταχύνουν την υλοποίηση των οικονομικών δράσεων. Στο δεύτερο τομέα, την γεωργία. Βλέπουμε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για να βεβαιωθούμε ότι οι εισαγωγικέ ε, ποσοστώσει δεν θα παραμείνουν αναξιοποιητέ για εμπορικού μόνον λόγου. Αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό, διότι σημαίνει περισσότερε ευκαιρίε για εξάπλωση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων. Επίση, συζητήσει γίνονται και για άλλου τομεί τη γεωργία. Ένα αφορά μια πρόταση να ασχοληθούμε με το πρόβλημα της αγοράς αποθήκευσης πόρων για την εγχώρια στήριξη και άλλο ένα άλλος ένας για τις δεσμεύσεις μας ως προς τις εξαγωγές και τον σχετικό ανταγωνισμό. Κάτι που απασχόλησε και τις συνομιλίες στην Τόχα και στους δύο, αυτού, δύο αυτούς τομείς είναι ακανθώδεις συζητήσεις και αναζητούμε μια πορεία προόδου Τίποτε δεν είναι βέβαιο, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και όσους ε, κάνουν τις προτάσεις και τις ανησυχίες όσων δυσκολεύονται να αποδεχτούν αυτές τις προτάσεις. Ένα τρίτο τομέας όπου αναμένουμε αποτελέσματα στον Παλί αφορά κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Όπω το να δημιουργηθεί μηχανισμό για την παρακολούθηση τη λειτουργία πολλών διατάξεων των κανόνων του ΠΟΕ για την μη διακριτική και προ προτιμησιακή μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών. Ελπίζουμε να περατώσουμε εδώ τι προτινόμενε αλλαγέ τη διατάξεις μα και επίση υπάρχει και σοβαρή πιθανότητα οι συμμετέχοντε να εγκρίνουν και μια δέσμη μέτρων για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε που να στοχεύει ειδικά αυτέ. Στο Μπαλί το φως των προβολέων θα πέσει και στην πρωτοβουλία του ΠΟΕ Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο. Ένα, θα έχουμε την τέταρτη έκθεση για το θέμα αυτό και την παρουσίασή της τον Ιούλιο φέτος στη Γενέβη, γιατί ως τώρα η εμπορική αυτή πρωτοβουλία μας έχει αποσπάσει σοβαρότατες υποσχέσεις από τις χώρες που αύξησαν σε 35 δις δολάρια το 2010 το 2% δηλαδή, σε 2% αύξηση τον προπολογισμό για τους σκοπούς αυτούς. 2% παραπάνω από όταν ξεκίνησε η όλη πρωτοβουλία. 6 δις δολάρια το 2011 λοιπόν, αποσπάσαμε γι' αυτό, δεν έχουμε ακόμη αριθμούς για το 2012, αλλά εδώ υπογραμμίζεται η σημασία της παρακολούθησης και της εξέμπρεσης πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση και την οικοδόμηση περαιτέρω δυνατοτήτων. Ολοκληρώνοντα τη σημερινή μου παρουσίαση, να θίξω δύο ακόμη ζητήματα. Οι πρόσφατε εξελίξει σε σχέση με τι περιφερειακέ εμπορικέ συμφωνίε πρώτον και το πώ συσχετίζονται με του πολυμερεί κανόνε του ΠΟΕ και το δεύτερο, η προσφατότερη έκθεση του Γενικού Διευθυντή Λαμή για το εμπορικό πάνελ. Ξέρω ότι θα τα συζητήσετε αυτά υπό το επόμενο σημείο τη σας διαταξή σα, αλλά να κάνω κάποια σχόλια και εγώ από την πλευρά μου. Πρώτα απ' όλα για τι περιφερειακέ εμπορικέ συμφωνίε. Είναι σαφέ έναντι των απογοητευτικών αποτελεσμάτων και τη βραδία προόδου τη πολυμερή διαπραγματεύση με τον κύριο τη Δόχα, οι περιφερειακέ εμπορικέ συμφωνίε έχουν αρχίσει να γίνονται ελκυστικοί, εναλλακτικοί. Βλέπουμε να υπάρχει εδώ κινητικότητα. Και διατλαντικό στο εμπόριο και στις σχέσεις Ασίας, ε, Ασίας Ειρηνικού, και βλέπουμε μια, ένα πολλαπλασιασμό των περιφερειακών συμφωνιών. Το θέμα ουδέποτε έπαψε να το σχόλιο των ΠΟΕ, διότι βεβαίω έχουμε περιφερειακέ εμπορικέ. Ε, ε, μάλλον μηχανισμό για τι περιφερειακέ εμπορικέ συμφωνίε, σύστημα κοινοποίηση και διαφάνεια για τι συμφωνίε αυτέ και πραγματικά η έκθεση, η εμβληματική έκθεση του ΠΟΕ για το εμπόριο του 2011 αφιωσίωσε ένα μεγάλο τμήμα στο θέμα αυτό. Και καταλήξαμε σε δύο γενικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, η αύξηση, ο πολλαπλασιασμό των συμφωνίων αυτών θα παραμένει μια τάση και για το εγγύ μέλλον. Και έπειτα, οι περισσότερε από τι συμφωνίε αυτέ ξεπερνούν τι αυστηρά παραγωγικέ πτυχέ ασχολούνται με τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση και ενσωμάτωση κανόνων, αριθμίσεων, προτύπων και πολιτικών επιλογών. Και αναφέρει η έκθεση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει πώς να ε, πάρουν πολυμερή ε, διάσταση οι περιφερειακές εξελίξεις. Για ανταγωνιστικά σήματα, λόγου χάρη. Θα πρέπει εδώ στις Βρυξέλλες να σκεφτούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη και άλλες μεγάλες οικονομίες όπως η Αμερική, ο Καναδάς και η Ιαπωνία για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέση εργασία φυσικά. Τέτοιε συμφωνίε πρέπει να αντιμετωπίζουν πραγματικού φραγμού που δυσκολεύουν το εμπόριο μεταξύ αυτών των χωρών. Όλο και περισσότερο τα εμπόδια αυτά μεταξύ αναπτυγμένων χωρών έχουν να κάνουν με μη δασμολογικού φραγμού και όχι δασμολογικού. Ρυθμίσει, κανόνε και πρότυπα. Θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε πραγματικά ωφέλη εδώ αν μπορούσαμε να άρουμε τέτοιου είδου φραγμού. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με λίγα λόγια για το πάνελ που ίδρυσε ο Γενικό Διευθυντή Λαμή για τα θέματα εμπορίου. Ο Γενικό Διευθυντή ε, δημιούργησε το πάνελ αυτό με 12 εξέχοντα μέλη που, δεν, που είναι ανεξάρτητοι από κράτη, εμπειρογνώμονε και αναλύουν τι τάσει του εμπορίου για τον 21ο αιώνα. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης αυτού του πάνελ που θα συζητήσετε κι εσείς αφορά την σύγκληση. Τη σύγκληση των εμπορικών καθεστώτων του χωρών που είναι μέλη του ΠΟΕ αντικατοπτρίζει δηλαδή την πρόοδο των εξελίξεων της, χώρα, της μιας χώρας προς την άλλη. Επίσης, τη σύγκριση των πολυμερών με τα διμερή συστήματα, το, συζήτηση, το σχολείο αυτό προηγουμένω, το αναφέρει και η έκθεση, ...την σύγκληση του εμπορίου με άλλου τομεί τη δημόσια πολιτική. Δηλαδή, αυτό που αναζητούμε είναι μεγαλύτερη συνέπεια στα μη δασμολογικά μέτρα αλλά και σύγκληση του εμπορίου με άλλες εγχώριε δημόσιε Καινοτομία, λόγω χάρη, ή κοινωνικές πολιτικές. Η έκθεση αυτή δεν δίνει απαντήσει Είναι μια απλή πρόσκληση για να συλλογιστούμε πώς ε, το αυριανό διεθνές σκηνικό θα μπορούσε να διαμορφωθεί, πώς θέλουμε να το ε, σχεδιάσουμε και τι ε, προσδοκούμε. Περιμένω λοιπόν και τη δική σας ενισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια, τις δικές σας απόψεις για την έκθεση αυτή και τις δικές σας εκτιμήσεις. Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω εδώ και πραγματικά είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας ή να ακούσω σχόλια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά να σας ακούσουμε. Τώρα προτείνω το σημείο για το μέλλον του εμπορίου. Να το δούμε κατόπιν. Και να ακούσουμε τώρα τον πρώτο ε, ομιλητή, τον Βραζιλιάνο βουλευτή. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία συμμετέχει σε συνάντηση της ε, Διευθυντικής Επιτροπής. Ε, πρόσφατα διοριστήκατε σε αυτή την Επιτροπή. Ήταν ε, μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή. Γιατί η Βραζιλία είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος της Διευθυντικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται έτσι κι από εκπροσώπους με γεωγραφική ε, κατανομή από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μας. Η Βραζιλία λοιπόν είναι ευπρόσδεκτη. Η Βραζιλία κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα του ΠΟΕ. Έχει πλέον νέες ευθύνες για το εμπόριο και πραγματικά ελπίζω να φτάσουν αυτά τα λόγια και στο Βραζιλιάνικο Κοινοβούλιο. Το γνωρίζω καλά γιατί έχω πάει μια-δυο φορέ ω εκεί. Κύριε Ούγκο Ναπολιάου, έχετε το λόγο. Ah, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην μιλήσω ε, για το νέο Γενικό Διευθυντή για πέντε λεπτά. Μου είπε ο κύριος Σεργέη όμως ότι θα έχω ευκαιρία για κάτι τέτοιο και αύριο. Καλά έχω καταλάβει. Να το σχολιάσω τώρα ή αύριο. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. No, it will be brief, you know, uh, Μπορώ να είμαι πολύ σύντομο. Ξέρετε, στη Βραζιλία μιλάμε πορτογαλικά έτσι κι αλλιώ. Μπορώ να μιλήσω αγγλικά. Αν θέλετε μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά, αλλά σε κάθε περίπτωση αγγλικά μιλάω. Και γαλλικά άμα χρειαστεί. Μιλάω κι εγώ, κάνω νοήματα. Uh, Εντάξει λοιπόν, μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά. Ε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι όλων των αγαπητών χωρών που εδώ εκπροσωπούνται. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να εκφράσω την χαρά μου για, την πρόσφατο, για τον πρόσφατο διορισμό του συμπατριώτη μας Ρομπέρτο Αζεβέντου ως Γενικού Διευθυντού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η επιλογή του κυρίου Αζεβέντου αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής και εξέτασης υποψηφίων απέκλεισε άλλους ε, υποψηφίους. Δηλαδή εδώ υπάρχουν δύο λόγοι να καμαρώνουν όλοι οι Βραζιλιάνοι. Πρώτον, ότι αναγνωρίστηκαν οι προσωπικές αρετές και οι επαγγελματικές αρετές του πρεσβευτού ε, Ρομπέρτου Αζεβέντου, του οποίου η μόρφωση και η παιδεία είναι ένα υπόδειγμα για το τι μπορεί να παράγει και να προσφέρει η χώρα μας στους τομείς της ε, εκπαίδευσης και της δημόσιας δίκησης. Έχει πτυχίο ε, πολυτεχνείου από το Πανεπιστήμιο της Μπραζίλια και με μετά την ε, είσοδό του στην διπλωματία και την ενασχόλησή του με τις διεθνείς μέσω του Ινστιτούτου Ρίου Μπράνκου απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικά προσόντα για την ε, εξάσκηση της διπλωματίας επί 15 χρόνια, 15 χρόνια συστηματικής εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρόκειται για έναν βαθύ γνώστη, όχι μόνο της εσωτερικής λειτουργίας του φορέα, του παγκόσμιου αυτού οργανισμού, αλλά γνώστη και των τεράστιων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορεί να παραμένει στη γραμμή της επικαιρότητα ο οργανισμός αυτός και να ανταποκριθεί στη δυναμική εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορούμε να καμαρώνουμε είναι γιατί διαπιστώνουμε ότι παρόλο που επηρεάστηκε από τις προσωπικές του και επαγγελματικές του αρετές η επιλογή του κυρίου Αζεβέντου, αυτή η ίδια επιλογή μπορεί να θεωρηθεί ύψη τη σημασία για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερος για τη Βραζιλία. Ιδίω το σημερινό ε, ε, οικονομικό σκηνικό διεθνώ. Και βεβαίως και από την ε, οπτική γωνία των πολυμερών διαπραγματεύσεων. Αυτή η επιλογή και άλλες γεωπολιτικές διευθετήσεις που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσμο σηματοδοτούν την ανάγκη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου να προσαρμοστεί. Να προσαρμοστεί σε απαιτήσει πολύ διαφορετικές από αυτές που γνωρίζαμε όταν ιδρύθηκε το 1995. Και αυτό για να αντικαταστήσει τη Γενική Συμφωνία για τους Δασμούς και το Εμπόριο, το ΓΑΤΣ, τη Συμφωνία GATS. Ο νέος ρόλος που έχουν αναλάβει και πρέπει να διαδραματίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, η καταπολέμηση του προστατευτισμού, οι, μάχες ε, συναλλαγματικές, με τη, όπως απηχήθηκαν στις συνομιλίες της Ντόχα και ως κίνητρο για την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου είναι βασικά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν έτσι ώστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου να ανακτήσει την πρωτοπορία, την πρώτη θέση που κατέχει με φυσικό τρόπο στο παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι θα μπορέσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας οικονομικής τάξης που να είναι δικαιότερη και πιο συμμετοχική. Χωρίς καμία αμφιβολία το καθήκον αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Κατά την άποψή μου όμως, ο πρέσβης Ρομπέρτου Αζεβέντου έχει τερα... α... α... πολλαπλές ικανότητες να αντιμετωπίσει, έχοντας ήδη αποδείξει ότι είναι ένας πολύ καλός διαπραγματευτής που πετυχαίνει συνενέσεις. Έτσι κι αλλιώς η διεθνής θεώρηση που έχει για τα πράγματα καθώς και η πείρα του ε, καλύπτουν ε, το σύνολο των χωρών του κόσμου, όχι μόνο τη γνώση της Βραζιλίας. Εύχομαι λοιπόν ο, να μπορέσει στα νέα του καθήκοντα να συμφιλειώσει τα διαφορετικά συμφέροντα των 159 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και θέλω να καταγραφεί με την ευκαιρία αυτή ε, η έκφραση των συγχαρητηρίων μου προς εκείνον για τη λαμπρή του αυτή νίκη και οι ευχές μου για κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την... Ευχαριστώ. Πώς ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον προσκεκλημένο μας τον αναπληρωτή, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ε, ζήτησε να σχολιάσει εν συντομία, ο κ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο εν είδη απάντησης. Ασφαλώς θα ήθελα να εκφράσω τη δέσμευση που όλοι όσοι εργαζόμαθα στον ΠΟΕ ε, Όλοι γνωρίζουμε τον κύριο Αζεβέδο πολύ καλά, τον πρέσβη κύριο Αζανέβο. Ε, ήταν πολλά χρόνια στη Γενέβη και προφανώς είναι κάποιος ιδιαίτερος ικανός με μία εις ε, γνώση του διεθνούς εμπορίου και του πολυμερού συστήματος. Και είμαστε υπερήφανοι για το σύστημα επιλογής το οποίο αναπτύχθηκε στον ΠΟΕ αυτή ήταν μια πολύ κανονική μετάβαση που έγινε με πολύ ανοιχτό τρόπο. Είχαμε εννέα υποψηφίους και ήταν μια διαδικασία της οποίας προηγήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις. Είχαμε μια ανοιχτή συνεδρίαση όπου παρουσιάστηκαν όλοι οι υποψήφοι και έκαναν τις παρουσιάσεις τους και έγινε ε, αξιοκρατικά μια σωστή επιλογή αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό σημείο. Εφόσον γίνεται γενικό Διευθυντή, βεβαίω αναλαμβάνει μια νέα ευθύνη. Είναι, κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερο ευπρόσδεκτο. Είναι ο πρώτος γενικός διευθυντής ε, του ΠΟΕ, από τη Λατινική Αμερική, μια περιοχή ζωτικής σημασίας με ε, ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το μολυμερές ε, σύστημα και αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι κινούμεθα προς ε, μια πιο ε, προς μια μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ε, μελών του ΠΟΕ. Όταν γίνεστε γενικός διευθυντής ενός οργανισμού όπως είναι ο ΠΟΕ, δεν είστε πλέον εθνικός εκπρόσωπος. Όλοι όταν μπαίνοντα στον ΠΟΕ γινόμαστε διεθνείς υπάλληλοι, δεν έχουμε ένα διαβατήριο αλλά πολλά. Και ο ρόλος του Γενικού Διευθυντού δεν μπορεί παρά να είναι επιτυχής εφόσον υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι σε θέση να πετύχει την συνένεση και να οδηγήσει τις χώρες προς κοινέ λύσεις. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ε, ε, ε, αναμένουμε με ανυπομονησία την, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Γιατί η Βραζιλία είναι γνωστή για την αυστηρή ε, εκπαίδευση των διπλωματών της. Εγώ ο ίδιος ήμουν διαπραγματεύτης στις Ηνωμένε Πολιτείες και είχα μια μακρά μαθητεία στη γραμματεία και έμαθα να είμαι σκληρός όπως η, πρώην κυβέρνη, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση και όλοι οι άλλοι και νομίζω ότι εσείς ε, έχετε μια αντίστοιχη εμπειρία. Θα φέρετε στη δουλειά αυτή τη δική σας ε, γνώση και εμπειρία του κόσμου και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές ε, δυνατότητες να, είστε να, είναι ένας πολύ καλός ε, διευθυντής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αζεβέδο ε, είχε εμφανιστεί εδώ στην Επιτροπή, υπήρξε μια ακρόαση και είχαμε όλη την δυνατότητα όχι μόνο να γίνουμε μάρτυρες των ε, μεγάλων του ικανοτήτων να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, αλλά και να αξιολογήσουμε τα προσόντα του. Και εγώ ε, ε, μετά την εκλογή του είχα την ευκαιρία να του διαβιβάσω τα προσωπικά, προσωπικά τα συγχαρητήριά μου για το διορισμό του ως Γενικού Διευθυντού του ΠΟΕ. βεβαίως είναι ιδιαίτερος κατάλληλος για το θέμα αυτό που αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στον ε, ΠΟΕ. Και τώρα θα θέλαμε να συζητήσουμε άλλου είδου ε, εξελίξεις. Η Κάθριν ε, Μπίρντερ από τους Φιλελευθέρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα περίμενα, περίμενα τους άλλους να μιλήσουν πρώτα. Λυπούμε γιατί περίμενα στην αίθουσα που ήμασταν το πρωί περιμένοντα να τελειώσει προηγούμενη συνεδρίαση και να ξεκινήσουμε Τέλο πάντων, έκανα λάθο, άργησα να έρθω. Θέλω να πω πάντω ότι με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που άκουσα, ιδίω τι απόψει σα σε ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση. Όπως γνωρίζετε, πολύ χρόνο και πολύ προσπάθεια έχουμε δαπανίσει ε, στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΣΑΚΕ για τις διαπραγματεύσεις μιας συμφωνίας εμπορικής, είπα. Ε, Συμφωνία Εμπορικής εταιρική Σχέσης. Ήταν δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις. γεωγραφικούς λόγους έχουμε ομαδοποιήσει κάποιες χώρες. Τελικά όμως καταλήξαμε σε ομάδες όπως ε, παραδείγματος χάρη η Σάντεκ, ε, η Νοτιοαφρικανική ή μάλλον η Ανατολικοαφρικανική κοινότητα και άλλες που ναι μην πρόκειται για ομάδες γεωγραφικές αλλά δεν είναι από οικονομικής πλευράς ομιγενείς, είναι πολύ Το Καμερούν τώρα βλέπουμε ότι θέλει να αποσπαστεί και να διαπραγματευτεί εκτός τη ομάδα στην οποία ανήκει. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Θα ήταν ίσως σκόπιμο, ε, δεν ξέρω στην Τόχα αν μπορεί να συζητηθεί το θέμα αυτό, αλλά εσείς πώς πιστεύετε ότι επί τόπου θα λειτουργήσει αυτό ιδίως με κάποιες από τις μικρότερες οικονομίες στην Ευρώπη, κάπως τα έχουμε καταφέρει ως περιφερειακό ε, οικονομικό μπλοκ, αλλά και πάλι υπάρχουν εντάσεις. Ξέρετε, κατάγομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει και εκεί ε, μεγάλη ένταση. Υπάρχουν εντάσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν μιλάμε λοιπόν για περιφερειοποίηση, θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο πιο ε, αναλυτικά στο θέμα αυτό. Πρόεδρος. Όσοι θέλουν το λόγο παρακαλώ να σηκώνουν τα χέρια τους. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι η ΣΚΑ. Η ΣΚΑ από την Ενωτική Συμμαχία. Λάθος πρόεδρε, στους πράσινους ανήκω, προς το παρόν τουλάχιστον. Να απαντήσω κάποια πράγματα σε σχέση με τον ΠΟΕ. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχει μια ευρέως δεδομένη αντίληψη, θα έλεγα, στην Ευρώπη ότι ο ρόλος του ΠΟΕ υποβαθμίζεται, μειώνεται τελευταία και ότι υπάρχει ανάγκη βαθιών μεταρρυθμίσεων. Πιστεύετε ότι αυτή η ανάγκη μεταρρυθμίσεων λαμβάνεται υπόψη από τη νέα ηγεσία, από τη γραμματεία και ούτω καθεξής. Μια τέτοια μεταρρύθμιση πώς θα οργανωθεί ως διαδικασία. Και ένα άλλο ερώτημα. Ποιε θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι οι βασικέ γραμμέ, οι βασικέ συνιστώσει τη μεταρρύθμιση. Δεύτερον, αναφερθήκατε ήδη στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ΗΠΑ, τι ε, συνομιλίε που έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν μα είπατε τι επιπτώσει θα είχε μια τέτοια συμφωνία για τον ΠΟΕ. Τι αντίκτυπο θα είχε Στι εργασίε του ΠΟΕ η ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας ε, εμπορικής μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, ε, τα τελευταία 12 χρόνια δεν προχωράμε πολύ στο θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Με τη νέα ηγεσία μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια πρόοδο. Πρόεδρος, τώρα εκ μέρους της Ενωτικής Συμμαχίας, ο Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ελπίζω η απουσία συντηρητικών από το ECR δηλαδή και το ΕΛΚΑ δεν δείχνει αδιαφορία για το ΠΟΕ και το εμπορικό σύστημα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ για την παρουσίασή του. Να ευχαριστήσω και τον Βραζιλιάνο πρέσβη που μας μίλησε για τις ε, πρόσφατες θετικές πολιτικές εξελίξεις, ε, την εκλογή δηλαδή ενός εκπροσώπου από τη Λατινική Αμερική στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Και βέβαια ε, ότι είπατε για τις προκλήσεις ε, που αυτό συνεπάγεται για το πολυμέρες εμπορικό σύστημα. Σε μια από τις ακροάσεις είχε πει ο κύριος Αζεβέντο ότι αυτό που κάνει ο ΠΟΕ και αυτό που δεν κάνει ο ΠΟΕ επηρεάζει γενικώ στον πλανήτη και ότι το σύστημα επίλυσης διαφορών ελπίζει να γίνει καλύτερο για τα φτωχότερα μέλη του ΠΟΕ και βέβαια εσείς μιλήσατε για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη γεωργία και τις ε, περιοχές του κόσμου που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τις αναπτυσσόμενες ενδεχομένες περιοχές. See that growing of βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό διμερών ε, συμφωνιών ε, σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Πώς ε, το εκτιμάτε και μάλιστα από μέλη του ΠΟΕ. Αυτό δεν παρεμποδίζει την ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης. Αν δηλαδή υπάρχουν συμφωνίες αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας, τι γίνεται με τους υπόλοιπους, τις άλλες χώρες ο νέος Γενικός Διευθυντής, έχετε κηρύξει ως στόχο την ενίσχυση του ΠΟΕ, γι' αυτό σας το λέω. Δεύτερον, αυτή την πρόκληση της κοινοβουλευτικοποίησης, αν μπορώ να την πω έτσι, του ΠΟΕ, πώς τη βλέπετε. Εμείς εδώ καθόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβόλιο, έχουμε διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους, εξοχότες... Ε, θέλουμε λοιπόν να μας πείτε κι εσείς ε, αυτό, πώς το βλέπετε το στοιχείο της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, δηλαδή της ένλυσης του ΠΟΕ. Ενισχύει, θα ενισχύσει το πολυμερές εμπορικό σύστημα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. από τους ε, Ευρωπαίους Ελεύθερους Δημοκράτες. Ο ΠΟΕ έχει πολλές επιτυχίες όσον αφορά την άρση των εμπορικών ε, φραγμών. Ήταν ε, πολύ δύσκολο να διαπιστώσω το βαθμό στον οποίο ε, οι φραγμοί έχουν μειωθεί. Αλλά όλοι συμφωνούμε στο ότι υπάρχει μια σημαντική απάλληψη των εμπορικών φραγμών. Άρα, ποια είναι τα σημαντικά περιφερειακά μπλοκ, εάν προστατεύονται από εμπορικούς ε, δασμούς και τελωνιακούς δασμούς. Ε, ποια είναι η σημασία αυτή, τον, η δική του σημασία των 21ο αιώνα. Θα ήθελα να μας κάνετε μια σχετική ανάλυση των περιφερειακών μπλοκ. Ο Ντέβιτ Μάρτιν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, η δική μου ερώτηση σχετίζεται με τις επιτυχίες του ΠΟΕ όσον αφορά την απελευθέρωση, όπως είπε το Αγμάρ. Εγώ είμαι υποστηρικτής του ΠΟΕ, αλλά ορισμένες φορές διαρωτάμε κατά πόσο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και το σύγχρονο μοντέλο του κόσμου. Τρία παραδείγματα. Σε αυτό το κοινοβούλιο πολλοί ε, ασχολήθηκαν με τα θέματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεπία του ατυχήματος στο Μπαγκλαντές. Ε, και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται παρκώς στον ΠΟΕ. Ε, το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την κοινωνική ευθύνη των εταιριών για τα ατυχήματα και στο επίπεδο των θυγατρικών τους και των προμηθευτών τους. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα και στη δική μου χώρα είναι η φοροδιαφυγή, το οποίο, η οποία αυξάνεται λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και καθώς αυξάνεται η παγκοσμιοποίηση η φοροδιαφυγή καθίσταται ευκολότερη και θεωρώ ότι ένας οργανισμός σαν τον ΠΟΕ φέρει κάποια ευθύνη ως προς την εξέβρεση κάποιων λύσεων για αυτό το φαινόμενο. Εάν ε, συνεχίζετε να δικαιολογείτε την απελευθέρωση, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η απελευθέρωση δεν ε, διαστρεβλώνει την ικανότητα των κυβερνήσεων να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες της. Και η τελευταία ερώτηση αφορά την ψηφιακή οικονομία και το πώς ε, αντιμετωπίζουμε κάποια αγαθά τα οποία δεν έχουν υλική ένυρη μορφή, αλλά ψηφιακή. Εσείς δεν κάνετε καμία διάκριση μεταξύ των δύο. Αλλά και αν δεν κάνετε εσείς αυτή τη διάκριση είναι διαφορετικά αυτά τα αγαθά και έχουν διαφορετικό, διαφορετικό αντίκτυπο. Και οι καταχρήσεις που προέρχονται από την ψηφιακή οικονομία θα πρέπει επίσης να γίνουν αντικείμενο έρευνας εκ μέρους του ΠΟΕ. Ωραία λοιπόν. Ε, για την ε, διευκόλυνση του εμπορίου. Ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει στο Μπάλι. Ε, αναφέρεται ο Πασκάλ Λαμί ότι έχει πει ότι οι προσδοκίες σε σχέση με τις συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου θα είναι ε, δεν θα είναι ε, πολύ ε, ουσιαστικές, πολύ υψηλέ, συγγνώμη. Αυτές οι προβλέψεις αναμένεται να βελτιωθούν. Έχει γίνει κάτι τις προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία ενδεχομένως για την διευκόλυνση του εμπορίου. Υπάρχουν τέτοιες βάσιμες ελπίδες. Ωραία. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για πραγματικά αυτό το ευρύ φάσμα των ερωτήσεων και θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να τις απαντήσω. Και νομίζω ότι ένα σημείο εκκίνησης ε, είναι ίσως να δώσουμε λίγο σάρκα και οστά σε αυτή τη συζήτηση εν σχέση με την ε, περιφερειοποίηση ε, και την απλούστευση όχι για το σύστημα του ΠΟΕ, αλλά για μια ευρύτερη πολυμερή συνεργασία και για την διεθνή οικονομία εν γέννη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης εδώ. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές από τις περιφερικές προσπάθειες οι οποίες γίνονται έχουν συμπεριληφθεί κατά τη σύσταση του ΠΟΕ. Έχουν ληφθεί υπόψη. Ε, στην αρχική ΓΚΑΤ ε, διατυπώσαμε κάποιους κανόνες οι οποίοι αναγνωρίζουν ακριβώς την ανάγκη των περιφερειών να ολοκληρωθούν ε, το ταχύτερο δυνατό ε, και ε, όχι βεβαίως στην παγκόσμια κοινότητα, αυτό είναι προφανές. Η ευρωπαϊκή κοινότητα και η ευρωπαϊκή κοινή αγορά και οι χώροι ελεύθερων συναλλαγών κλπ ε, ενέχουν ε, κάποιους ε, κανόνες και την αναγνώριση ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εμφανίζει μια συνοχή με τις βασικές αρχές των μη διακρίσεων παγκοσμίω. Η μείωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών δασμών γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά γίνεται, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ γιατί ε, το να δημιουργεί μια εσωτερική περιφερειακή συνοχή ε, εις βάρος των εξωτερικών εταίρων δεν έχει, δεν έχει νόημα. Όλες οι πολυμερείς ε, συμφωνίες είναι φύση ε, έχουν ε, από τη φύση τους αυτή τη μορφή. Ε, αλλά αυτό δεν μας απομακρύνει από την ανάγκη να πρέπει κανείς να πληρεί τις προϋποθέσεις, τους βασικούς όρους, να υπάρχει μια ίση μεταχείριση βάσει των κανόνων του ΠΟΕ και όπως αυτή που υπάρχει και προς τους εξωτερικούς εταίρους. Και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το πρωτομισιακό σύστημα, αλλά όπως είπε ένας ομιλητής, όσο περισσότερο γίνονται διαπραγματεύσεις για τα προτιμησιακά συστήματα, τόσο λιγότερο σημαντικά γίνεται. Δηλαδή τελικά υπονομεύονται οι προτιμήσεις του προηγούμενου καθεστώτος μέσω, ενός νέου, μέσω διαπραγμάτευσης ενός νέου καθεστώτος οι περιφέρειες είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές και ε, δεν θα και θα πρέπει να πληρούν εξίσου τους ε, κανόνες όπως και οι άλλοι προμηθευτές. Τώρα έχουμε περίπου 300 ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ε, μεταξύ περιφερειών, οι οποίες έχουν αναφερθεί στους δικούς μας μηχανισμούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι σχολιαστές αναφέρονται σε αυτούς και το σημαντικό θέμα εδώ είναι πόσο επιπρόσθετος άχθος ε, κομίζει αυτή η πολυπλοκότητα των ε, διαφορετικών ε, συμφωνιών επί τη βάση διαφορετικών κανόνων αντί για την προσπάθεια να ενταχθούν σε ένα πολυμερές σύστημα. Και το ερώτημα που οποίο γύρεται για τον ΠΟΕ αφορά την σταθεροποίηση των πλεονεκτημάτων που ενέχει το πολυμερές ε, σύστημα. Και αυτό με βγει στο ερώτημα το οποίο τέθηκε σε σχέση με την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον ε, ΠΟΕ. Κατά πόσο μειώνεται η σημασία του ΠΟΕ ή όχι. Εγώ θα το διατύπωνα ως εξής. Ε, παρά όλες αυτές τις ε, διμερείς περιφερειακές συμφωνίες, οι μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο διέπονται από τους κανόνες του ΠΟΕ. αυτό ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή το εμπόριο με τις ε, ΗΠΑ βασίζεται στους κανόνες του ΠΟΕ. Το ίδιο και για το εμπόριο με την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και πολλές άλλες μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Ε, ωστόσο παρόλα αυτά και ε, παρά την ε, επικέντρωσή μας σε αυτού του είδους συμφωνίες, το πολυμερές ε, σύστημα είναι η μόνη προσφυγή που έχουν πάρα πολλές χώρες για να εξασφαλίσουν ότι οι εταίροι τους σέβονται τις ίδιες αρχές των μη διακρίσεων. Βασικές αρχές όπως η εθνική αντιμετώπιση υπάρχουν λίγοι που μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζονται εθνικές αρχές διεθνείς συμφωνίες. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει ένα, μια αρκετά σύνθετη επικάλυψη της πολυμερούς ε, προσέγγισης με όλες ε, τις άλλες τις υπόλοιπες διευθετήσεις. Παρ' όλα αυτά η πολυμερής προσέγγιση διατηρεί τη σημασία της. Δεν νομίζουμε ότι έχει ευθύνη και αν δείτε τις διαμάχες, τις διανέξεις που προσφεύγουν στον ΠΟΕ ε, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η ισχύς και η αξιοπιστία του ΠΟΕ γιατί πολλές ε, υποθέσεις τελικά ε, καταλήγουν στο μηχανισμό, στο όργανο διατησίας και διευθέτηση των διαφορών του ΠΟΕ. Τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες μιας ε, μεγάλης διμερούς ε, διαθέτησης. Αν δούμε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, διαπραγματευτούν μια συμφωνία ελεύθερων οικονομικών ε, συναλλαγών. Θεωρώ πραγματικά ότι αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση στο πολυμερές σύστημα. Ελπίζω αυτή η επίπτωση να είναι πραγματικά θετική, αλλά να δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κάποιος... Ε, εγώ δεν ζηλεύω την, το έργο των διαπραγματευτών ε, εδώ. Εάν ε, αυτό συμβεί, θα επηρεάσει το προσανατολ... τους προσανατολισμούς μας εντός του ΠΟΕ. Ε, κατά πόσο υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών που έχουμε συμφωνήσει με την ΣΥΠΑ και τους στόχους, τους κανόνες του ΠΟΕ. Ή αυτό θα οθήσει ορισμένες χώρες να διαπραγματευτούν ε, το δικό τους ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διαπραγματεύσεις με πολλούς άλλους εταίρους, για παράδειγμα τη Λατινική Αμερική, για τη σύναψη συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου και βεβαίως αυτό θα έχει μια μακροπρόθεσμη επίπτωση στο, ε, ε, στην πολυμερή προσέγγιση. Ένα ερώτημα τέθηκε σε σχέση με τους κανόνες του ΠΟΕ και με το κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη του τις ε, ουσιαστικές μεταβολές οι οποίες λαμβάνουν χώρα ε, και κατά πόσο διατηρούν το επίπεδο εναρμόνισης. Και θεωρώ ότι εάν ε, δούμε τι γίνεται στο εμπορικό περιβάλλον, εδώ ο ΠΟΕ έχει εξελιχθεί σε πολλά θέματα. Υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση της ανάγκης για ύπαρξη συνοχής μεταξύ, για παράδειγμα, εμπορικών και, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών. Ένα από τα, ένας από τους στόχους της Δόχα ήταν υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ ε, ΠΟΕ και διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Οι κλιματικές μεταβολές, εάν ε, μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε μια διεθνή περιβαλλοντική σύμβαση, δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι θα πρέπει να φτάσει στον ε, ΠΟΑ μια τέτοια συμφωνία. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ κυβερνήσεων, όχι διαπραγμάτευση στον ΠΟΕ. Αλλά ο ΠΟΕ θα πρέπει τη στιγμή εκείνη να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα έχει κάτι τέτοιο στους εμπορικούς ε, κανόνες. Ένα από τα πράγματα τα οποία θα χρειαστούμε καθώς ε, αναπτύσσουμε τον βαθμό συνοχής με περιβαλλοντικά θέματα είναι ακριβώς αυτή η συνοχή μεταξύ περιβαλλοντικών και εμπορικών ε, κανόνων. Τώρα, η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι βουλευτές. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω εν γέννη είναι ότι ο ΠΟΕ ασφαλώς έχει γίνει ένα θεσμικό όργανο το οποίο λαμβάνει όλο και περισσότερο υπόψη ε, το, την πολιτική όφηση το, κάτω από πολλές οπτικές γωνίες. Ε, τα μέλη του ΠΟΕ είναι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται μεταξύ τους, αλλά από την άλλη έχουμε όλο και περισσότερο, όχι μόνο την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση να έχουμε μία αλληλεπίδραση μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων του ΠΟΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς ε, και της μη κυβερνητική ε, κοινότητας και τους βουλευτές. Εάν δείτε το Δημόσιο Φόρουμ, το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο στη Γενέβη, εκεί έχουμε μεγάλη συμμετοχή βουλευτών και γίνονται πολύ έντονες ε, συζητήσεις για τα θέματα αυτά θέσατε κάποια ερωτήματα για, σε σχέση με τη φοροδιαφυγή και υποθέτω ότι όντως θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο πλατιά την δημοσιονομική ρύθμιση και τον αντίκτυπό της στο διεθνές ε, εμπόριο. Ε, ε, είναι, πράγματι υπάρχουν πολύ λίγοι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα τη φορολογία ε, και γίνονται συζητήσεις κατά πόσο οι φόροι επί των εξαγωγών ε, βρίσκονται σε συμφωνία, είναι συμβατές με τη συμφωνία. Ε, υπάρχει λοιπόν μια σχετική αντιπαράθεση, συζήτηση με το πω, αλλά η φορολόγηση δεν είναι το πεδίο που ο ΠΟΕ έχει διαδραματίσει ιστορικά καθοριστικό ρόλο. Ιστορικά ήταν ε, μία δέσμη συμφωνιών που σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με την ε, συναλλαγές ε, αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, και δεν νομίζω ότι ε, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ενδεδειγμένο φόρουμ για θέματα συζήτηση μεταξύ υπουργών οικονομικών σε σχέση με τη φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα, η G20 ε, και τα θέματα τα οποία συζητούν δείχνουν την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και σε άλλους τομείς πέραν των καθαρά οικονομικών συναλλαγών, δηλαδή των τελωνιακών δασμών κλπ. Ενδεχομένως ορισμένοι ε, θέλουν να δουν πώς εμείς ε, είμαστε πετυχημένοι όσον αφορά τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου συστήματος κανόνων και ενός μηχανισμού διευθέτησης των διαφορών. Και ίσως θα ήθελαν να μεταφέρουν το σύστημα αυτό σε, σε άλλα πεδία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει πολύς ε, χρόνος ε, ότου οι κυβερνήσεις ε, είναι πρόθυμες να υπαχθούν σε ένα διεθνές σύστημα φορολόγησης. Και αυτό με οδηγεί στο να θέσω το ζήτημα της ψυχιακής οικονομίας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν το προσφέρει ο ΠΟΕ. Μιλάμε για ιδιωτικού ε, εμπλεκομένους φορείς ε, που όμως πράγματι είπαν ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή προχωρούμε προς αυτή την ψηφιακή οικονομία. Οι συναλλαγές ε, αγαθά και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν. Στον ΠΟΕ το έχουμε συζητήσει για πολύ καιρό ιδίω για το ηλεκτρονικό εμπόριο συγκεκριμένα που είχαμε μία ε, συζήτηση και εκεί πολλά βέβαια ε, ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία τα συζητήσαμε. Ένα μείζον ζήτημα είναι ποιοι είναι εθνικοί περιορισμοί και πολιτικές σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε σχέση με την φορολόγηση των ελόγων συναλλαγών. Όμως, όλο και περισσότερο θα συζητείτε και το θέμα της ε, συνάφειας των κανόνων του για, τα, ε, για την επίλυση των διαφόρων. Δεν το συζητήσαμε, αλλά φαντάζομαι ότι στην ε, Συμφωνία περί θα τα συζητήσουμε πληρέστερα όλα αυτά τα ζητήματα. Τέλος, ό,τι αφορά την πρόγνωση που κάνατε για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, θα ήθελα να πω ότι προχωρούμε πολύ καλά προς επιτευξή συμφωνία στον Παλί για την ε, διευκόλυνση των συναλλαγών. Σίγουρα υπάρχουν πολλά κανθόδη στήματα, αυτό είναι αλήθεια. Είναι έντονη η διαπραγματεύσεις, σίγουρα, και ίσως το καλύτερο για μένα ως ε, αξιωματούχο του ΠΟΕ είναι να είμαι διπλωματικός ή καλός διπλωμάτης. Τι θα πει αυτό, είχε πει κάποιος ε, ένας καλός διπλωμάτης είναι αυτός που σκέφτεται δύο φορές πριν μιλήσει. Και επειδή υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν θα ήθελα να πάρω κάποια, κάποιο το μέρος εδώ και να τοποθετηθώ, αλλά ελπίζω στον Παλί να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γιατί αυτό θα είναι και ένα μήνυμα, μια ένδειξη ότι μπορούμε ακόμη να τα καταφέρνουμε στο επίπεδο του ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρο, σας περάσουμε τώρα στο σημείο 23. Μένουμε ε, στο θέμα του παγκοσμίου εμπορίου και το θέμα μας είναι το μέλλον του εμπορίου, οι προκλήσεις της σύγκλησης. Αυτό το έγγραφο θα συζητήσουμε που σας δείχνω ουσιαστικά. Πρόκειται για μια έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για το μέλλον του εμπορίου. Την ομάδα αυτή τη συγκάλεσε πέρυσι, το 2012 δηλαδή, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, Πασκάλ Λαμή. «24 Απριλίου δημοσιεύτηκε έκθεση, πρόσφατα δηλαδή. Αντίγραφα της έκθεσης μπορείτε να τα βρείτε στο βάθος έθουσας και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Στόχος μας εδώ σήμερα είναι να έχουμε μια πρώτη συζήτηση της έκθεσης αυτής. Οι προκλήσεις της σύγκλησης λοιπόν. Έχουμε καλέσει τον κύριο Ράινχαρτ Κουίκ. Συνεργάτη του Προέδρου της Business Europe. Συνομοσπονδίας ε, των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. πρόεδρος, ε, ε, ο πρόεδρος Θούμαν ήταν και μέλος αυτής της ομάδας. Ο κύριος Σουίκ είναι και πρόεδρος ε, της ομάδας Εργασία της Business Europe για τον ΠΟΕ. Θα γίνει πρώτα η παρουσίαση. Αν δεν μπορείτε να μείνετε για τη συζήτηση, μάλιστα. Καλά, θα μας παρουσιάσετε λοιπόν το θέμα και εν συνεχεία η κυρία Γιόργενσεν, τακτική θαμώνας των συνεδριάσεών μας, θα πάρει τώρα να μας πει τα υπόλοιπα. Πού είναι, πού είναι ο προσκεκλημένος μας κύριος Κουίκ, Κύριε Ράινχαρτ Κουίκ, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της έκθεσης για το μέλλον του εμπορίου. Ο κύριος Θιούμαν, μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω σήμερα, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί. Η έκθεση είναι μια ενδιαφέρουσα σύνοψη των προκλήσεων που εντοπίζει σήμερα το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Άκουσα ορισμένο ε, ε, παρεμβάσεις ε, στην προηγούμενη συζήτηση που νομίζω ότι αντανακλούν το ότι ορισμένα ζητήματα από αυτά που και εσείς συζητήσατε μας ενδιαφέρουν και τα έχουμε περιλάβει και στην έκθεσή μας. Η έκθεση αυτή υπερβαίνει βέβαια τα σημερινά προβλήματα Δεν θα βρείτε πάντως κάποιες ε, συστάσεις για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα, αλλά πιο πολύ τα συστημικά ε, συγκεκριμένα ζητήματα ε, εξετάζουμε. Λαμβάνουμε υπόψη τις νέες εμπορικές πραγματικότητες και ιδίως τις παγκόσμιες αξίες και τις αλλαγές. Global Value Change είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση ε, και θα πρέπει να θέσουμε το εξή ερώτημα. Οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες πώς θα πρέπει να στηρίζουν την, ε, τις, ε, τις παγκόσμιες αλυσίδες αυτές, Global Value Chains. Έχουμε διάφορα θέματα, πρότυπα, κανόνες, επενδύσεις, υπηρεσίε μη δασμολογικά εμπόδια και ούτω καθεξής. Για τις ε, αλυσίδες αυτές λοιπόν θα πρέπει να δούμε σε ζητήματα όπως είναι η κατάργηση των δασμών για τα ενδιάμεσα προϊόντα. Αν με επιτρέπετε μία προσωπική άποψη, η απελευθέρωση των ε, δασμών για περιβαλλοντικά προϊόντα, για παράδειγμα, δεν ανταποκρίνεται νομίζω σε μια απελευθέρωση στην παγκόσμια αλυσίδα αξιών. Πόσα προϊόντα χρειάζονται για παράδειγμα για την παραγωγή ενός ηλιακού συλλέκτη ή μιας ε, τουρμπίνας. Φυσικά και απελευθέρωση είναι καλή εν γέννη, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο να επηρέαζε την όλη παραγωγική αλυσίδα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης, που νομίζω ότι δίνουν κάποια χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το παγκόσμιο εμπόριο, τα ωφέλη της ε, απελευθέρωσης του εμπορίου και το πώς βλέπουμε το εμπόριο γενικότερα μέσα στο διεθνέ πλαίσιο. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα θέμα σημαντικό, του μη δασμολογικού φραγμούς. Υπάρχουν ε, δασμοί, ε, όσο υπάρχουν και συνεχίζουν να, να παρακολουθούν δηλαδή, την ανταλλαγή προϊόντων, βέβαια υπάρχει μία μείωσή τους, ιδίως σε σχέση με την ε, περιοριστική δράση που έχουν οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Ο ΠΟΕ συμφωνεί με αυτά, αλλά θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο για να διαμορφώσει το θεματολόγιο του εμπορικό για τον 21ο αιώνα. Το θέμα αυτό που αναφέρω το έχετε συζητήσει κι εσείς και μάλιστα το συζήτησα και στην προηγούμενη συζήτηση. Πώς θα βρεθεί λοιπόν η ισορροπία, πώς θα έχουμε κίνητρα δημόσιας πολιτικής και πώς θα τα εξορροπήσουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης, ε, κατά την άποψή μου. Ένα άλλο παράδειγμα. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες στον ΠΟΕ για τον ανταγωνισμό. Επιδοτήσεις για πρώτες ύλες δούμε της ενέργειας, για παράδειγμα. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε αμυντικά εμπορικά μέτρα στην προσπάθεια να έχουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο Business Euro πάντοτε υποστηρίζαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των δασμολογικών φραγμών στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων της ΔΟΧ. Γιατί θα ήταν ίσως αποτελεσματικό μέτρο για να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και να δώσουμε λύσεις χωρίς να χρειάζεται να, παρα... Ε, να προσφεύγουμε συνεχώς τον μηχανισμό επίλυσης διαφόρων του θα ήταν εθελοντικό ο μηχανισμό αυτός για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων τα οποία προκαλούνται από την επιβολή με δασμολογικών μέτρων. Θα ήθελα τώρα εν συντομή να σας παρουσιάσω το μέλλον του ΠΟΕ, το τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της έκθεσης. Αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχει στήριξη για τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης εθνικής ε, προτίμησης της, ε, της μεταχείρισης μάλλον του πλέον ε, προνομιακού εταίρου κτλ. Θα πρέπει πιστεύω να παραμείνουν αυτές οι βασικές αρχές στο ΜΠΟΕ. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται συνετικά οι αποφάσεις. Για λόγους διαφάνειας πάντως τα μέλη του ΠΟΕ που είναι αντίθετα στις αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να δίνουν τριτολογημένη ε, τους άποψη. Έρχομαι στις προτιμιασιακές εμπορικές συμφωνίες. Βλέπουμε ότι πιο πολύ ε, η πλάστιγκα κλείνει προς τις διμερές, διμερείς και όχι πολυμερείς συμφωνίες. Όμως, έχουμε κάποια θέματα. Can be considered Οι συμφωνίες αυτές όμως θα μπορούσαν να είναι θετικές οι πλειονομερείς αυτές εμπορικές συμφωνίες. Είπαμε για τη συμφωνία ελευθέρωση των αλλαγών με τη Αυτό θα μπορούσε να προωθήσει την απελευθέρωση και τη ρυθμιστική συνεργασία. Ή θα προωθήσει και το εμπόριο με τρίτες χώρες. Όχι μόνο μεταξύ ΙΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστική όμως αυτή η συμφωνία. Είδαμε, για παράδειγμα, την απόφαση και της Ιαπωνίας πρόσφατα να προχωρήσει ο TPP. Εμένα δεν με ε, ανησυχεί το μέλλον του ΠΟΕ ιδιαίτερα. Εγώ πιστεύω ότι θα μεγαλώσει η σημασία του. Γιατί? Το TPP και το TPIP θα είναι πραγματικά ε, γνήσιες εμπορικές συμφωνίες του αυτό αποτελεί και ένα πρότυπο, ένα μοτίβο στο οποίο πάνω θα πατήσουν άλλες ε, συμφωνίες. Δημιουργεί απόκληση η σύναψη ε, τέτοιων συμφωνιών Μήπως μετά υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να εξαλείψουμε. Αν πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, μόνο μέσω του ΠΟΕ μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης αν όλες οι προσεγγίσεις της Συμφωνίας Ελεύθερων Σταγών αποτύχουν, που ελπίζω να μην συμβεί αυτό, αλλά αν συμβεί, θα πρέπει πάλι να πάμε στη Γενέβη. Επομένως, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γενέβη, αγαπητοί φίλοι. Επίσης, στην έκθεση περιλαμβάνονται και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ρόλο του ΠΟΕ στο μέλλον. Θα επικεντρωθώ σε τέσσερις περιορισμούς των εξαγωγών, τον έφερε ο κύριος Γέξα. Πρέπει ο ΠΟΕ να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ε, περιορισμών των εξαγωγών. Απαγορεύονται οι ποσοστώσεις. Οι φόροι όμως εξαγωγές δεν απαγορεύονται. Τι κάνουμε επίσης με τα ε, συστήματα διπλής τιμολόγησης για τους φυσικούς πόρους, για παράδειγμα η πολιτική ανταγωνισμού επίσης. Δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατικών επιχειρήσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό μας ανησυχεί. Θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση διεθνών κανόν ανταγωνισμού. Θα πρέπει αυτή η κανόνες να εφαρμόζονται και σε κράτη. Εγώ μπορώ να σκεφτώ μη ανταγωνιστικές ε, συμπεριφορές κάποιων κρατών. Επενδύσεις ήταν στην ατζέντα, αλλά δυστυχώς βγήκε από τις επανατεύσεις της Ντόχα. Αλλά αν δείτε αυτή την παγκόσμια λυσίδα αξιών, θα καταλάβετε πόσο σημαντικές θα είναι οι συμφωνίες για τις επενδύσεις. Και ίσως θα έπρεπε να είχαμε μια πολυμερή ε, επενδυτική συμφωνία. Τέλος, ο ρόλος της γραμματείας. Ε, ξεκάθαρα στην έκθεση αναφέρεται ότι η γραμματεία του ΠΟΕ θα πρέπει να έχει ισχυρότερο ρόλο να διαδραματίσει. Ε, βέβαια, ε, όπως πάντοτε μας έλεγαν, ε, είναι μια οργάνωση η οποία πιο πολύ κατευθύνεται από τα μέλη της και κάποιες φορές υπήρξαν κάποια κράτη ήταν εχθρικά σε κάποιες εξελίξεις. Αν δείτε όμως προτιμησιακές συμφωνίες, κάποιες από αυτές εγώ δεν θεωρώ ότι συνάδουν τους κανόνες του ΠΟΕ, Κανείς όμως ε, δεν προσβάλλει τις συμφωνίες αυτές ε, στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Γιατί μήπως η γραμματεία του ΠΟΕ θα έπρεπε να έχει το ρόλο να προσβάλλει τέτοιες συμφωνίες ως θεματοφύλακας, για παράδειγμα, της συνθήκης. Οι Ευρωπαίοι νομίζω εύκολα θα μπορούσαν να το δεχθούν αυτό. Τέλος, ε, Μιλάμε στην έκθεση για τη σύγκληση εμπορικών καθεστώτων των κρατών μελών του ΠΟΕ μεταξύ πολυμερού συστήματος ε, διμερών και πολυμερών πρωτοβουλειών, μεταξύ εθνικών πολιτικών και άλλων. Πολύ σύντομη ήταν η παρουσίαση αυτή. Μια έκθεση πολύ μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση. Thank ε, βεβαίως, η παρουσίαση της, η έκθεση είναι ιδιαίτερως περιεκτική, περιλαμβάνει 40-50 σελίδες θα έλεγα. Αυτή όμως ήταν πολύ καλή σύνοψη η κυρία Γιώργενσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή μου να παραστώ εδώ γιατί θεωρούμε η εργασία που γίνεται στο IPU για το πολυμερές σύστημα ε, ιδιαίτερος ε, ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εξαιρετική έκθεση που έχει προετοιμάσει το Πόνελ, αλλά επίσης ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, κ. Λαμή, που έχει ξεκινήσει αυτό το έργο και υπάρχει μια, είναι πολύ ισορροπημένη προσέγγιση και ε, είναι μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση σε σχέση με το ρόλο του διεθνούς εμπορίου και της ε, πολυμερούς προσέγγισης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε στο πολυμερές ε, σύστημα για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση του εμπορίου και θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ενίσχυσης αυτού του πυλώνα. Το πολυμερές σύστημα είναι δημόσιο αγαθό και όλα τα μέλη θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πόρους τους για να το ενισχύσουν και είναι σημαντικό σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία σημαντικών προκλήσεων ε, κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι εισηγητές. Ο ΠΟΕ προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια για περαιτέρω εξέλιξη του προβληματισμού και μας δίνει μια σημαντική ανάλυση για τις ε, μεταβολές στο πολυμερές σύστημα και διατυπώνεται κάποια συστάσεις για την ανάληψη δράσεων και που διαιρούνται σε τέσσερα στρατηγικά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στην ε, παρουσίαση. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω στο πρώτο από αυτά τα ερωτήματα το οποίο είναι πώς θα ε, προχωρήσουμε στην, ε, πώς θα εξελίξουμε την ατζέντα της Δόχα. Ο λόγος που θέλουμε να, θέλω να επικεντρωθούμε εδώ είναι το γεγονό ότι θεωρούμε κεντρική σημασία για την οργάνωση του διεθνού εμπορίου. Η ενδεχόμενη ελοκλήρωση του γύρου τη ε, Ντόχα είναι προπόθεση για την ενίσχυση του ΠΟΕ και θα καλύψει η επίλυσή της και άλλα θέματα του ΠΟΕ. Ε, χωρίς την ολοκλήρωση αυτής της ατζέντα υπάρχει ο κίνδυνος, το πολυμερές σύστημα και ο ΠΟΕ τελικά να υπονομευθούν από άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις που τελικά θα υποσκάψουν το πολυμερές σύστημα και τις βασικές του αρχές. Συμφωνούμε ότι τέτοιες προσεγγίσεις έχουν ένα τεράστιο δυναμικό, αλλά απουσιάζει η παγκόσμια διάσταση την οποία παρέχει ο ΠΟΕ. Το πάνελ ε, κάνει κάποιες ε, συστάσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της ατζέντα της Δόχα, αλλά ε, τονίζει την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την αμοιβαιότητα και την ευελιξία, η οποία σέβεται τις διάφορες πραγματικότητες των χωρών που βρίσκονται σε, διάφορο διαφορετικό επίπεδο εξέλιξης. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αμοιβαιότητας και ευελιξίας, κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν και είναι ακρογωνιαίες λήθος της πολιτικής μας. Αυτό το ζήτημα της ευελιξίας και διαφοροποιημένης ε, αμοιβαιότητας είναι παρόν ε, σε άλλους τομείς ε, όπου επιζητούμε ακριβώς αυτή την ευελιξία. Εάν αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, θα ησυχάσουν οι ανησυχίε όλων μας και όπω το έθεσε ο Πασκάλ εμείς στο παρελθόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο οι αναδυόμενες οικονομίες είναι ε, ε, πλούσιε ε, οικονομίε με πολλού φτωχού ή φτωχέ χώρε με λιγότερου φτωχού. Ε, και όλα αυτά βεβαίως σχετίζονται με, το, με την πολυμερή προσέγγιση και νέα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ΠΟΕ και να υπάρξει και μια αναθεώρηση του συστήματος. Ε, ε, και αυτό μας φέρνει στη βασική η ερώτηση πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις πολυμερείς ε, συζητήσεις. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος τα μέλη του ΠΟΕ να μην είναι σε θέση να συμφωνήσουν ε, στα βασικά αποτελέσματα της διευπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο αυτού του έτους. Από την άποψη της επιχειρηματικής ε, κοινότητας σε πολλά μέρη του κόσμου, ο οργανισμός ε, αρχίζει να καταραίει σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες που άρχισαν να αναδύονται και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ανησυχητικό ότι το γεγονός ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ φαίνεται να παίζουν κάποια παιχνίδια ελιγμών, τακτικών ελιγμών, και αυτή τη στιγμή στη Γενέβη υπάρχει πρόοδος για την διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά το θέμα αυτό γίνεται όμοιρος ορισμένων χωρών μελών που θέλουν να προωθήσουν άλλα θέματα ε, που και ενδεχομένως τον τρόπο αυτό υποσκάπτει τη δυνατότητα του ΠΟΕ να πετύχει μια συμφωνία το Δεκέμβριο. Ε, έχει, υπάρχει δέσμευση τα μέλη να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις στους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί κάποιοι πρόεδροι, ούτως ώστε να δουν οι βάσεις για την περαιτέρω εργασία. Ανησυχούμε ότι, ότι τα μέλη του ΠΟΕ δεν, μπορούν, δεν θα μπορέσουν να πετύχουν μια συμφωνία σε μια πραγματικά απλή και χρήσιμη διευκόλυνση του εμπορίου αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, πώς θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε πιο δύσκολα θέματα όπως είναι η πρόσβαση ε, στην αγορά, η απελευθέρωση των υπηρεσιών και η γεωργική παραγωγή. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω τώρα εν συντομία τις περιφερειακές συμφωνίες ε, και τη δική μας δέσμευση στις πολυμερείς συμφωνίες. ξεκινήσαμε μια μεγάλη κλίμακα διμερών συμφωνιών, οι οποίες βεβαίως ενέχουν κάποιους ε, κινδύνους, αλλά κάνουμε μια συνεχή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και βλέπουμε σαν μέσο να προετοιμάσουμε τις πολυμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ αποστέλλοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα της βούλησής μας να ανοίξουμε τις αγορές σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και να ασχοληθούμε με σύνθετα ρυθμιστικά θέματα, μπορούμε να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη και αυτό είναι το βασικό σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από την παρούσα μας ε, δέσμευση. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο τέτοιε είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να βρουν ένα κοινό παρανομαστή σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να διαδραματίσει το δικό του ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Σήμερα η παγκόσμια παραγωγή ε, κάνουν τον ε, ΠΟΕ ως πολυμερή πυλώνα ακόμα πιο σημαντικό. Υπό το πλαίσιο αυτό συμφωνούμε με το συμπέρασμα του πάνελ ότι τα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να εστιάσουν τις, ε, την προσοχή του στα υφιστάμενα θέματα στην παρούσα ατζέντα ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι ξεκάθαρος, θα πρέπει να έχουμε μια πετυχημένη διυπουργική συνδιάσκεψη ως αναγκαία προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της ατζέντα της Δόχα και περαιτέρω εργασία σε άλλους τομείς που είναι σημαντικές για την ατζέντα της Δόχα. Αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και στην προσπάθεια να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα. από την IPU. Έχουμε συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν τώρα στους προσκεκλημένους από την IPU. Ο Χέλμουντ Σόλτς είναι ο πρώτος ομιλητής από την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί νομίζω ότι είναι για όλους μας ξεκάθαρο με την παρουσίαση της έκθεσης αυτής που ουσιαστικά προετοιμάζει και τη συζήτηση για την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Και θα το συζητήσουμε μέχρι το Δεκέμβριο πολλές φορές το όλο θέμα. Θα έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πιο εντατικά για όλα αυτά τα θέματα που πραγματεύεται αυτή η έκθεση. Να σχολιάσω καταρχάς τις σελίδες 6 και 12, όπου αναφέρεται το ζήτημα του Aid for Trade, βοήθεια το εμπόριο. Υπάρχει πρόκληση και των επενδύσεων για το εμπόριο. Μήπως λοιπόν θα ήταν δυνατόν να μας εξηγήσετε λίγο πιο αναλυτικά πώς θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, πώς μπορεί να ενταχθεί και στη δομή του ΠΟΕΔΕΦΤΕΡΟΝ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και από τον πρώτο γύρο να συσχετίζουμε τις προκλήσεις του πολυμερούς εμπορικού συστήματος σε ό,τι αφορά το TPP και τα λοιπά. 25 25-26. Έχουμε μια περιγραφή των δασμολογικών μέτρων που επηρεάζουν όλο και περισσότερο το εμπόριο. Θα ήθελα να θέσω ένα πρόβλημα που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο ότι το εμπόριο θα πρέπει να δει και τη γενικότερη, μάλλον θα πρέπει να λάβει υπόψη τους και τις γενικότερες οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Δηλαδή, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χώρες μέλη, σε ό,τι το εμπόριο, ποια είναι η σχέση με την οικονομική πολιτική που ακολουθούν υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση με τις δημόσιες πολιτικές. Jones Act είναι ένα παράδειγμα αυτό. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα είναι πρόβλημα να ξεπεράσουμε αυτό το από καιρό ισχύον νομοθέτημα τον είπα. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα πολυμερές σύστημα που θα λειτουργεί. Πώς επηρεάζει λοιπόν ε, αυτό το σύστημα τις δημόσιες πολιτικές των κρατών μελών του ΠΟΕ. Και λέει επίσης έκδοση ότι μπορεί εμπόριο να βελτιώσει την κατάσταση της ε, ισότητας σε Σελίδα 30. Μειώνονται οι τιμές στην χώρια οικονομία με το εμπόριο. Συμβάλλει το εμπόριο στη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των μελών. Τελικά, οικονομικές, ε, οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών είναι κάτι συγκεκριμένο, απτό. Μπορούμε να βρούμε κοινούς ε, συμπεφωνημένους κανόνες για την ενίσχυση, την επανενίσχυση του παγκόσμιου συστήματο. Και βέβαια το μείζον θέμα είναι η γεωργία και εδώ βλέπω και στην παρουσίαση να υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Υπάρχουν χάρη στη σελίδα 5 των συμπερασμάτων και επειδή μετά ακολουθεί και στη σελίδα 35 μια πιο αναλυτική περιγραφή και βλέπουμε κάποιες αντιφάσεις, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Uh, Ευχαριστώ από τους πράσινους η κυρία, Κέ... Κέλλερ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτής της ενδιαφέρουσας έκθεσης. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις και θέλω να ακούσω για τις επενδύσεις για το εμπόριο, investment for trade. Πάντως, ε, σίγουρα στα σημεία σύγκλησης της έκθεσης συμφωνούμε ότι πρέπει να ε, υπάρξει πολυμερής αντιμετώπιση των ε, περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει να ασχοληθούμε με το πολυμερές πλαίσιο και την ένταξη σε αυτό και των υπηρεσιών. Πάντως, η Συμφωνία για τις Κυβερνητικές Προμήθειες δεν βρήκε πολλούς σύμφωνους πέρα των χωρών που αποφάσισαν να διαπραγματευτούν αυτές τις για έξω. Υπάρχει λοιπόν κανένα επιχείρημα που να μας λέει ότι θα συμφωνήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες με αυτήν την τάση σύγκλησης. Και υπό την ίδια σκοπιά για τα θέματα της Σιγκαπούρης που οδήγησαν και στην αποτυχία της διπουργικής του Κανκούν το 2003. Μα πιέζουν εδώ οι αναπτυσσόμενε χώρε για διεθνεί κανόνε ανταγωνισμού και για πολυμερεί επενδυτικέ συμφωνίε. Τι σα έχει κάνει να αλλάξετε γνώμη και να προτείνετε εκ νέου την εξέταση αυτών των θεμάτων. Θέματα που ήταν αμφιλεγόμενα και στο επίπεδο του ΠΟΕ και που δεν τα στήριξαν οι επισόμενες χώρες. Έχει αλλάξει αυτό πρόσφατα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Ε, Ο από Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Τον Οκτώβριο του 2010 στο Στρασβούργο με πλειοψηφία 2 τρίτων ε, είχαμε πάρει μια απόφαση στο θέμα των διαπραγματεύσεων με τη Σούρ που λέει ότι καλείται η Επιτροπή τις ε, γεωργικές εισαγωγές προς την Ευρώπη, να τις επιτρέψει μόνον εφόσον ε, ισχύει η προστασία, η τήρηση των ε, προδιαγραφών για το περιβάλλον και σεβασμού των ζώων και προστασίας της υγείας. Και αυτή την απόφαση στήριξαν όλες οι πολιτικές ομάδες και θα με ενδιαφέρει να μας πείτε κατά πόσο τηρεί η Κομισιόν αυτές τις προδιαγραφές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία για την προστασία των φυτών και στη συνέχεια να επιτρέπουμε να επιτρέπουμε την εισαγωγή προϊόντων ε, που, από χώρες όπου χρησιμοποιούνται μαζικά κάποια ε, ε, κάποιες, ε, κάποια δημοκτόνα πολύ βλαβερά. Uh, Ο κύριος Ρινάλντι από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή, διότι πιστεύω ότι μια σειρά συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θετικά. Θα ήθελα να θέσω όμως κάποιες ερωτήσεις. Γιατί. Γιατί προκειμένου να επιτύχουμε, πιστεύω, σε διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, είτε διμερείς είτε πολυμερείς, πρέπει να έχουμε και κάποιο είδου σύγκληση μεταξύ των εταίρων μέσα από μέτρα που θα αποφασιστούν και θα υλοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο. Διερωτώ με, τι είδους μελέτη τι είδους αποτίμηση μπορεί να υπάρχει για αυτό το τομέα ιδιαιτέρως. Πιστεύω ότι με περισσότερο εμπόριο μπορούμε να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, αρκεί να υπάρχει ένα υγιές προλογικό σύστημα σε διεθνές επίπεδο, το οποίο να στοχεύει στην ανακατανομή των ε, εισοδημάτων που αποκομίζει το εμπόριο. Αυτό ε, προϋποθέτω ότι θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, κάτι που αποτελεί πάντοτε πειρασμό. Όπου υπάρχουν εμπορικέ δραστηριότητε, δημόσιε προμήθειε, προμήθειε και το καθεξή. Ξέρουμε εδώ τέτοια παραδείγματα. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια ρητή μνήμα τη καταπολέμηση τη διαφθορά, που δεν είναι όμω αρμοδιότητα του ΠΟΕ και που μέσω εθνικών αρχών επιλύεται με βάση την επικουρικότητα. Αλλά είναι απαραίτητο για να γίνει επιτυχέστερο το εμπόριο. Και σε ένα τρίτο επίπεδο πρέπει να συγκινήσουμε και την κοινή γνώμη τις μη κυβερνητικές ε, ε, οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις ενώσεις καταναλωτών, εργοδοτών, εργαζομένων και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες σε ένα χώρα αλλά πρέπει και κάποιε φορές να δούμε τι γίνεται και με τα εθνικά κοινοβούλια, που είτε συμμετέχουν πλήρως, είτε είναι ένας περιθωριακός συνομιλητής, ανάλογα με τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι η προσπάθεια σύγκλησης πρέπει να συμπεριλάβει ε, όλα αυτά τα στοιχεία της διεθνού πολιτικής, τα οποία πρέπει να ε, ισχύσουν ταυτόχρονα για να υπάρξει πραγματικά επιτυχία. Πρόεδρος, κύριε Χάρισον. Πρόεδρε, αυτό που είπε ο κύριος Γέρσα για τους βουλευτές με σημάδεψε. Εδώ έχουμε ευρωβουλευτές, αλλά και συναδέλφους από κοινοβούλια ή από την κοινοβουλευτική συνέλευση καλύτερα του ΠΟΕ. Εγώ αναφέρθηκα σε ένα βήμα της έκθεσης της επισκόπησης που μιλάει για το πλησίασμα των συνομιλητών μας, των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιοι από τους παρεμβαίνοντες έχουν συγκεκριμένες ιδέες βλέποντα τα πώς αυτά μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά. Ξέρουμε παραδείγματα από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ, από συνδικαλιστικές οργανώσεις, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τι γίνεται με την εξέταση εμπορικών θεμάτων. Που είναι βεβαίως κάτι σημαντικό για την κάθε μια από τις χώρες μας ξεχωριστά. Στη Βουλή των Λόρδων πρόσφατα αναλάβαμε μια δέσμευση ενώπιον με κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων προκειμένου να εξετάσουμε τους στόχους μας για τη διπουργική. Ελπίζω αυτό να γίνει και αλλού. Ξέρω ότι εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο ε, συζητάτε τα θέματα αυτά με μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Ντεχούχτη ήταν εδώ το πρωί και ήταν ακριβώς ένα μέρος της όλης συζήτησης. Πρόεδρος, Βεβαίως και οι δικές μας εμπειρίες είναι εδώ πολύτιμες και προσδεκτές. Η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ε, είναι μέρος της ε, διαδικασίας μας, όπως προβλέπετε για το διαφορμένο διάλογο, αλλά είχαμε μια έντονη συζήτηση με τον Επιτρόπο Ντεχού, επιτρόπο που είναι αποφορτισμένο με τα θέματα εμπορίου. Επιτρέψτε μου τώρα να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Να είμαι ειλικρινής. Επογοητεύτηκα λιγάκι από την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων στην έκθεση αυτή. Και έχω την εξή ερώτηση. Αυτή η, η έκθεση είναι καρπός ε, της άσκησης αυτοεγκράτειας από τα μέλη της Διευθυντικής Επιτροπής, η έλλειψη προτάσεων δηλαδή, ή το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και δεν υπάρχει μια συνταγή και συμφωνία στη συνταγή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ποια ήταν η αντίδραση στην έκθεση αυτή, εάν υπήρξε, στους διαδρόμους του ΠΟΕ. Έχετε καμιά είδηση σχετικά. Και τώρα να δώσω το λόγο και πάλι σε συναδέλφους. Ποιος ζητά το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, μπορείτε να συστηθείτε. Για τα πρακτικά. Μισελ Ναζάλα από την Ιορδανία. Η έκθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως σωστά είπατε. Τίτλους θεμάτων, αλλά τίποτε το συγκεκριμένο, ωστόσο. Ε, βλέποντας τι εμπειρίες έχουμε από την Ιορδανία και πώς είναι η κατάσταση με γενοτήρια, γειτονικέ χώρε που έχουν φθηνότερη ε, στη στην ενέργεια ή ε, στο ενεργειακό κόστο και στα προϊόντα του και στο εργατικό δυναμικό ε, υπάρχει άμεσο αντίκτυπο στο εμπόριο. Και υπάρχουν χώρε που μα εμποδίζουν στην ελεύθερη διακίνηση πορευμάτων. Κάτι που του επιτρέπει να ελέγχουν τη διακίνηση των Ιορδανικών προϊόντων. Είμαστε από τι πρώτε χώρε που υπογράψαμε και προσχωρήσαμε στον ΠΟΕ. Έχουμε πολλά προβλήματα λοιπόν στην περιφερειά μα και πολλά, πολλές δυσκολίες. Αυτά όλα θίγονται με τίτλους, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό που να προτείνεται. Πιστεύουμε ότι οι βιομηχανοποιημένες χώρες έχουν υποφεληθεί πολύ περισσότερο από την ε, συμφωνία του ΠΟΕ της Ντόχα από ό,τι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ιορδανία. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για, για θέματα που πραγματικά καίνε τις, ε, είναι καυτά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, περισσότερο από ό,τι για τις εκβιομηχανισμένες. Πρόεδρος, νομίζω ότι κύριε Ναζάλ αυτό το πάνελ δυστυχώς δεν θα ετοιμάσει δεύτερη έκθεση εγκαίρως. Ας ε, περάσουμε και πάλι στον κατάλογο των αγορητών. Ο κύριος έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω η πρώτη ερώτηση, το Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο. Εάν σκεφτείτε ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία εμπορικών διευκολύσεων, θα έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς οι μελλοντικές επενδύσεις μπορούν να οργανωθούν ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από ένα περιβάλλον ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων ταχύτερα, διασυνοριακά. Αυτό βοηθείται και υποβοηθείται και από την ίδια τη δομή του ΠΟΕ. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατανόησα την ερώτηση για τα μη δασμολογικά μέτρα. Νομίζω και το είπε ο κ. πολύ σωστά, ότι ο ΠΟΕ δίνει μεγάλο χώρο πολιτικό ε, για την κατάρτιση εθνικών πολιτικών, ιδίω ω προ την εμπορική ευθυγράμμιση και την επίλυση εμπορικών διαφορών. Θέματα που έχουν τεθεί επανειλημμένω στον ΠΟΕ. Το αν πάντοτε η ποιότητα είναι υψηλότερη χάρη στην ε, παρέμβαση του ΠΟΕ, εντάξει, μπορείτε να αμφιβάλλετε, αλλά το θέμα είναι το εξή. Οι φραγμοί, όταν αρθούν, επιτρέπουν μεγαλύτερη απελευθέρωση, άνοιγμα και τελικά ευημερία. Το αν υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία για τη γεωργία και τις πολιτικές επιλογές σχετικά με τη γεωργία. Στην έκθεση αναφέρεται ότι υπάρχουν ε, δυνατότητες πολιτικών ελιγμών ώστε να μην πληγεί ο ανταγωνισμός. Στο επόμενο στις επόμενες ερωτήσεις τώρα. Για τις επενδύσεις. Τι έχει αλλάξει. Νομίζω αν κοιτάξει κανείς τι έγινε τα τελευταία 50 χρόνια, ένα πράγμα που έχει σίγουρα αλλάξει, και αυτό αναφέρεται στην έκθεση, είναι οι διεθνείς τιμές. Πώς εμπορευόμαστε πλέον τις μέρες μας. Εάν θέλουμε να, να επηρεάσουμε τις ε, τιμές διεθνώς και τα προϊόντα που παράγονται διεθνώς, δεν με και εγώ ίδιο, δεν χρειάζεται μια επενδυτική συμφωνία. Οι χώρε που θέλουν να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν στην αλυσίδα των ε, τιμών διεθνώς, στην παραγωγική αλυσίδα, δεν χρειάζονται μια διεθνή επενδυτική συμφωνία που να την έχουν ε, εγκρίνει και να την έχουν κυρώσει, ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από την αλυσίδα αυτή. Εάν δεν έχουν υπογράψει, πώ το ωφεληθούν. Αυτό λέω και εγώ στον εαυτό μου. Κάποιε αλλαγέ τι είδαμε τα τελευταία 15 χρόνια και ο ΠΟΕ τι απηχεί. Το 2001 ακόμα όμω δεν τι είχε λάβει επαρκώ υπόψη του. Τώρα, για την ερώτηση που τέθηκε για την διαφθορά και την διαφάνεια. Όσο πιο πολλές κυβερνήσεις έχουμε, τόσο καλύτερες εμπορικές σχέσεις διαμορφώνονται. Και όσο καλύτερη διακυβέρνηση έχουμε, τόσο περισσότερο πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Βέβαια, το δύσκολο είναι να πετύχουμε σύγκληση σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Αυτό ήταν ένα θέμα που ανέκαθεν μας προβλημάτιζε. Τι πολιτικούς ελιγμούς, τι περιθώριο πολιτικών ελιγμών ε, μπορούμε να αφήσουμε και πώς ένα συγκεκριμένο εμπορικό μέτρο, μια συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να αντιφάσει και με εμπορικούς κανόνες. Εδώ προσπαθούμε να βρούμε ακριβώς τη σωστή ισορροπία. Και η έκθεση διασφαλίζει και προστατεύει το περιθώριο πολιτικών ελιγμών. Αν δείτε τι έγινε με την επίλυση διαφορών και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, 20 χρόνια πριν ένα τέτοιο πάνελ δεν θα μπορούσε να έχει διοργανωθεί. Θα ήταν ασύμβατο με τον ΠΟΕ. Νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια πάνελ. Τέτοιες εξελίξεις ακριβώς για να προβλέπεται και ο πολιτικός χώρος για τις απαραίτητους έλεγμους. Δεν μπορώ να σχολιάσω για τη συμμετοχή των ε, κοινοβουλευτικών. Απλώς ξέρω ότι γίνεται με το κοινοβουλευτικό φόρουμ του ΠΟΕ και βρίσκω ότι είναι χρήσιμη εμπειρία. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο και έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσε συζητήσει με τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερομένων. Βεβαίω υπάρχει τάση επιχειρηματίε να μένουν μεταξύ του και οι πρόσωποι των κυβερνητικών οργανώσεων το ίδιο, αλλά τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είχαμε χρήσιμε και παραγωγικέ συζητήσει. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν είναι συγκεκριμένο, πρέπει ο ΠΟΕ να το πάρει και να το αξιοποιήσει. Πάντω αυτό με φέρνει και στη δική σα ερώτηση, Πρόεδρε. Λέτε ότι απογοητευτήκατε που δεν έχουμε συγκεκριμένε χειροπιαστέ προτάσει. Αν διαβάσετε προσεκτικά την έκθεση, θα δείτε ότι οι προτάσει υπάρχουν. σω να μην είναι συγκεκριμένε. Αν ήταν όμω πιο χειροπιαστέ, θα μα επέκριναν. Θα μα λιντσάριζαν και θα μα έλεγαν ότι να πάλι, συγκεκριμένε προτάσει που κανεί δεν τι υλοποιεί. Και έχετε δίκιο. Πού είναι η πολιτική βούληση να προχωρήσει ο ΠΟΕ, να προχωρήσει πιο μπροστά Υπάρχει πολιτική βούληση σε αυτή τη φάση. Ναι, όντως ασκηθήκαμε στην αυτοεγκράτεια εδώ, στην αυτοσυγκράτηση, γιατί μπορεί εσάς να μην σας φαίνεται αρκετό, αλλά εάν δείτε που βρισκόμαστε στις ε, διεθνείς συνομιλίες, τι λέει η έκθεση. Λέει ότι υπάρχουν πολλά θέματα όπου οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν μετά την τόχα. Στη φάση μετά την τόχα. Και είναι σημαντικά θέματα αυτά. Οι εξαγωγικοί περιορισμοί, οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες. Είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε και να πάρουν σχήμα. Αλλά εάν μια τέτοια έκθεση μπορούσε να κάνει προτάσεις, πώς θα γινόταν τα μέλη να αποφασίζουν εάν υπάρχει πολιτικό περιθώριο και δυνατότητα να γίνουν διαπραγματεύσεις και να βρεθούν συμφωνίες για τέτοια θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Κυρία Γιώργινσεν, αναφέρατε ότι κάποιες χώρες εκβιάζουν τις καταστάσεις προκειμένου να πετύχουν παράλληλους στόχους τους. Μπορείτε να τις κατονομάσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα προτιμούσα όχι, αλλά ελπίζω όλες οι χώρες να ακολουθήσουμε μια πιο επικοδομητική προσέγγιση στη Γενέβη, ώστε για τον ΠΟΕ και για την επίλυση των διαφορών να έχουμε θετικές εξελίξεις. Δεν είμαι από τις συντάκτες της έκθεσης, άρα θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα όσα αφορούν την Κομισιόν και μετά θα κάνω κάποια πιο γενικά σχόλια για ορισμένα άλλα ζητήματα. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν για την ρύθμιση σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά, φυτογειονομικά, ε, το σχετικό κανονισμό για την ασφάλεια των τροφίμων μας. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα πληρέστατο πολύ καλό πλαίσιο υγειονομικής φυτογειονομικής νομοθεσίας που φυσικά εφαρμόζεται και στις εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται πλήρως. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι φυσικά και εφαρμόζουμε τον κανονισμό μας και όπου χρειάζεται θα προβούμε και σε περαιτέρω ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια των, και την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα που αφορούσαν τον αντίκτυπο του εμπορίου, στην ισότητα, την ανάπτυξη των χωρών. Πάνω σε αυτό θα σας παραπέμψω στο έγγραφο του Προέδρου Μπαρόσο που το επέβαλε το Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων αναφερόταν και σε αυτό το θέμα, επενθυμίζοντας τη σημασία των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων και ότι θα πρέπει τα κράτη να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως όλα τα ωφέλη του πολυμερού συστήματος. Επίσης, ε, υπήρξε η κριτική ότι είναι πολύ γενικόλογες ε, ορισμένες από τις συστάσεις της έκθεσης. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό, η οποία αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφορών των ΠΟΕ, την ανάγκη για ευελιξία, τις ευθύνες των χωρών σχέση με τα άλλα κράτη κτλ. Και νομίζω ότι εκεί ε, σε αυτή την σύσταση για την ευελιξία υπήρχε ε, ένα επίπεδο μεγαλύτερης λεπτομέρειας και ακρίβειας. Δεν ήταν τόσο γενικόλογο όπως άλλα αυτό το κομμάτι, αυτό το σκέλος. Τώρα, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις σημαντικές αλλαγές ε, που έχουν επισυμβεί στην παγκόσμια οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία, ίσως και παραπάνω και πρέπει να δούμε πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν ε, το πολυμερές εμπορικό σύστημα, πώς μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στη Γενέβη και στον τρόπο της οργάνωσής μας. Είπατε, με ρωτήσατε για την παρουσίαση ε, της έκθεσης στη Γενέβη, τι λεγόταν στους διαδρόμους κτλ. Όταν ε, υποβλήθηκε στον ΠΟΗ έκθεση υπήρχαν ε, πράγματι κάποια μέλη τα οποία αναγνώρισαν ότι μεταξύ των ε, εμπειρογνωμονών υπήρχαν σημαντικές διαφορές. Γι' αυτό και χρειάστηκε να διατυπωθούν γενικόλογες συστάσεις επί σειράς θεμάτων, εκτός που παραλαμβάνω της ευελιξίας και της διαφοροποίησης. Πάνω σε αυτά ήθελα να σχολιάσω, αλλά αν υπάρχουν και άλλα ερωτήματα προς την Κομισιόν, ευχαριστώ να επανέλθω. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνουμε τη συζήτηση επί του σημείου 23. Να ευχαριστήσω τα μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΠΟΕ που ήταν παρόντα για τη συζήτηση των δύο αυτών σήμερα της διάταξης. Μπορείτε να παραμείνετε και για τα υπόλοιπα σημεία τη διάταξη, ε, ακόμη και αν αυτά δεν αφορούν τον ΠΟΕ. Αλλιώ, ε, αν φύγετε, σα υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε μια συνάντηση στι 10. Ελάτε γύρω στις 9 και 4 για να ξεκινήσουμε ε, ακριβώς την ώρα μας στις 10 γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε στη συνεδρίαση της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής του Steering Committee. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο σημείο 20. See you tomorrow then.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 όσοι αποχωρούν να το πράξουν ησύχως ε, και τάχιστα. Για να προχωρήσουν παρακαλώ. Okay. Next item again. Item 20. Σημείο 20 λοιπόν. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή ΕΜΒΗ, που είναι καθήλυνα αρμόδια για το νομοθετικό αυτό ζήτημα που αφορά την τροποποίηση τη οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και τη οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ. Η Χωσέφα Αντρέ είναι η εισηγητριά μα και θα συζητήσουμε αυτή τη φορά τροπολογίε των συναδέλφων προ το σχέδιο γνωμοδότηση Your help, please. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βοηθήστε με. Ησυχία παρακαλώ. Η Χωσέφα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται για γνωμοδότηση, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ΕΜΒΗ αλλά όπως νομίζω ότι είχαμε σχολιάσει και σε μια ε, συνεδρία της ομάδας εργασίας, ε, πρόκειται για την πρώτη ε, γνωμοδότηση. Εμείς δηλαδή ουσιαστικά θα ανοίξουμε κάπως το θέμα. Πρόκειται για την ποιότητα των καυσίμων λοιπόν, και τις ανανεώσιμες πηγές. 103 τροπολογίες, αν και λίγες, κατατέθηκαν θέτουν λοιπόν υπόψη μας τη σημασία της γνωμοδότησης αλλά και της έκθεσης. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ένα εξ αυτών είναι η αναγνώριση ε, του υπολογισμού. Το είχαμε συζητήσει, δεν είναι τέλειο. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε να είναι αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα τα στοιχεία και να μπορούμε να τα υπερασπιστούμε σε περίπτωση προσφυγής. Επίσης για τον υπολογισμό του ε, διοξιδίου του άνθρακα από την προθεσμία που τίθεται ε, είναι καλό ε, στοιχείο, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κριτήρια βιωσιμότητας και για τη δεύτερη και όχι μόνο για την πρώτη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά. Το μοντέλο δεν νομίζουμε ότι είναι ε, παρκώς όριμο για να δρομολογηθεί αμέσως, γιατί θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος για να έχουμε κάποια ευελιξία Τότε φορά το ΚΑΠ είχαμε μία τροπολογία να έχουμε την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες στον υπολογισμό του 10%. Θα τροποποιούσε βέβαια αυτό το μοντέλο της Κομισιόν και αυτό θα επηρέαζε και την αγορά. Αν διατηρήσουμε αυτό το κριτήριο υπολογισμού ίσως να μην δοθούν επαρκώς κίνητρα για τα βιοκαύσιμα της δεύτερης γενιάς. Αυτός όμως είναι ο στόχος της έκθεσης, να προωθήσουμε τα καύσιμα δεύτερης γενιάς. Θέλουμε λοιπόν να καταθέσουμε μια τροπολογία για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης ενδιαφέροντα είναι αυτά που λέγονται για την μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα των εθνικών συστημάτων βιωσιμότητας. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Δεν ξέρουμε πού μπαίνει αυτό στην οδηγία αυτή. Είναι αρμοδιότητα των κρατών. Πού πρέπει να το εντάξουμε. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ίσως μας το διευκρινίσει η Κομισιόν όταν λάβει το λόγο. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Η έκθεση είναι αρκετά τεχνική και πολύπλοκη. Έγιναν αρκετές τεχνικές συναντήσεις και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με βάση αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν Σίγουρα όμως να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί σας είπα ότι υπήρξαν ζητήματα που δημιουργήθηκαν και σίγουρα έχουν προκύψει και προσδοκίες μετά την πρόταση της Κομισιόν. Για το κάτω μοντέλο σας θέλω να ξέρω και για τη βιωσιμότητα του μοντέλου σας. Είναι σημαντικά για να προχωρήσουμε. Yes, 100 uh, amendments Το δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Ακούσουμε τώρα τους ε, σκιώδες. Η Ελίζαβεθ Κιώστιγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ε, ευχαριστούμε πολύ ε, την εισηγήτρια για τα εισαγωγικά της λόγια. Και εγώ χαιρετίζω το γεγονό στην πρώτη τεχνική συνάντηση μεταξύ σκιωδών ε, αποκρισταλώθηκαν κάποια σημεία όπου, ε, των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια της βιωσιμότητας. Θεωρώ ότι εδώ θα είναι εφικτό εντός της, ε, ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων να υπάρξει μια προσέγγιση και να εξευρεθούν κάποιες λύσεις. Τα πιο προβληματικά πεδία αναφέρθηκαν ήδη από την εισηγήτρια και είναι ασφαλώς το μοντέλο υπολογισμού προσμέτρησης και η πολλαπλή μέτρηση. Ήδη εδώ κάναμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό και πολλές επιτροπές έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ακόμα και η Επιτροπή ήδη σε ορισμένες της ε, γνωμοδοτήσεις ε, ε, είπε ότι αυτό το μοντέλο υπολογισμού ε, είναι σφαλμένο, δεν είναι δεδειγμένο και δεν ε, οδηγεί ε, σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Και θα ήθελα να πω, δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν λέει ότι ναι, δεν είναι τέλειο, αλλά χρειάζεται μια βάση υπολογισμού. Έχει δίκιο, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να συμφωνήσουμε με ένα μη αξιόπιστο σύστημα υπολογισμού, γιατί με τον τρόπο αυτό θα προκαλέσουμε περισσότερες ε, ζημίες. Και υπάρχει μια μελέτη από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου, το οποίο λέει ότι αυτό το μοντέλο ε, ε υπόκειται σε πολλές διακυμάνσεις ανάλογα με την ε, χρήση διαφόρων παραγόντων ε, προσμέτρησης της ε, αξίας ε, της καύσης των, ορυκτών, των τιμών για τα ορυκτά καύσιμα, τιμών καύση για τα ορυκτά καύσιμα. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε σε αυτή τη βάση να καταλήξουμε σε πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή βασιζόμενοι σε ένα μη αξιόπιστο μοντέλο. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι εδώ και το δεύτερο σημείο αφορά τις πολλαπλές ε, μετρήσεις. Και το ε, θέμα αυτό τέθηκε από την εισηγήτρια και είναι πολιτικά δημοφιλές με απλά λόγια να διαχωρίσω τα πράγματα σε άσπρο μαύρο. Αλλά ιδιαίτερα ε, στον τομέα παραγωγής ενέργειας χρειαζόμαστε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση και μια τεχνητή το να δημιουργεί μια τεχνητή στάθμιση μεταξύ διαφόρων ομάδων ε, ε, ισοδυναμεί με το να μιλάμε σε άσπρο μαύρο για καλά και κακά βιοκαύσιμα. Έχουμε διάφορες γενναίες, ε, πιο πραγματικά και πιο συμβατικά βιοκαύσιμα και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα καύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά όχι με τέτοιου είδους ε, διαφοροποίησεις, ε, διαχωρισμούς μάλλον μεταξύ άσπρου, μαύρου, καλού, κακού ε, τα πρόβατα και τα ερήφια. Και νομίζω ότι τι, σημαίνει για τα βιοκαύσιμα όταν τα μετράμε πολλαπλά. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει στο αντίθετο αν, έχουμε μόνο 25%, αν υπάρχουν μόνο 25% ενός ορισμένου καυσίμου, ε, ενώ για άλλο καύσιμο ε, ε, έχουμε 100%, τότε στην περίπτωση αυτή έχουμε μια απώλεια της τάξης του 75% και κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο και ούτε και οικονομικό και θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό να ζημιωθούν και νομίζω ότι θα έπρεπε να δείξουμε κάποια σύνεση και να εξετάσουμε τι είναι αυτό που μακροπρόθεσμα ε, ε, τι σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα για την οικονομία της Ευρώπης και για το ισοζύγιο πληρωμών στον τομέα των καυσίμων. Ε, το ισοζύγιο στον τομέα των καυσίμων. νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό τελικά θα ευνοηθεί μια περαιτέρω εξάρτηση και ίσως στον τομέα αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις τεχνικές λεπτομέρειες και να έρθουμε σε πολιτικά σωστές ε, λύσεις. Επόμενη μιλήτρια είναι η Κάθριν Μπίρντεν από το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή έκθεση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει αυξάνουσα σημασία λόγω των απρόβλεπτων επιπτώσεων. Θέλαμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άθρακα και θεωρήσαμε ότι βρήκαμε μια καλή λύση, αλλά στην πραγματικότητα υπήρξαν πολλοί έξυπνοι, οι οποίοι είναι πιο έξυπνοι από εμά ξύπνοι οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν περισσότερα χρήματα με ενδιαφέροντες ε, τρόπους και το οποίο τελικά οδήγησε σε αλλαγές της χρήσης γης, κάτι το οποίο δεν είχαμε προγραμματίσει αρχικά. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν καθέσει πολλές τροπολογίες και νομίζω, αλλά νομίζω το έχουμε προσεγγίσει με ένα επικοδομητικό τρόπο. Ιδιαίτερα σε αυτή την επιτροπή είχαμε ε, αντιστοίχως περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες και ορισμένες φορές ε, ε, τελικά ασχοληθήκαμε με τα πορικά ζητήματα, που να πούμε ναι ή όχι. Αλλά στη δική μου τροπολογία 24 ζητούμε να υπάρχει μια πολύ πλήρους έκθεση σε αυτή την Επιτροπή. Ε, λογοδοσία. Ε, όσον αφορά την κυριότητα γης στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ένα τροματικά δυσχερές ε, πρόβλημα. Δεν είναι ζήτημα που αφορά το εμπόριο, αλλά όταν μιλούμε για αυτό το θέμα της αλλαγής των χρήσεων γης, συνδέεται με το γεγονός ότι πολλά πράγματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν ε, μια... δεν υπάρχει μια κατάλληλη δομή αναγνώρισης της κυριότητας της ε, γης. Και ε, ορισμένοι ε, παίρνουν, υφαρπάζουν τη γη από τους προύχοντες των χωριών, ζυομιώνοντας τρομακτικά τις ντόπιες κοινότητες. Έχουμε συζητήσει ε, ε, για μακρόν στην Επιτροπή αυτή τη σχέση μεταξύ εμπορίου και περιβάλλοντος. Ε, στη Κολομβία, όπου είχαμε πάει, ασκήσαμε τεράστιες πιέσεις και φαίνεται οι προσπάθειες αυτές να καρποφόρησαν και ε, γη που είχε υφαρπαγή ε, πεστράφει στους ε, πραγματικούς κατόχους της. Ένα από τους άλλους, ένα από τα άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι το ζήτημα της διαφάνειας. Και αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι θα δω και καιρό και πιέζουμε ε, γιατί αυτό αφορά τόσο τις καλλιέργειες όσο και την ε, δασοκομεία και τις εξορρεκτικές δραστηριότητες. Η, διαφορ... η διαφάνεια είναι ένας τρόπος όπου μπορούν ε, μέσω της οποίας μπορεί να, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους οι, οι αυτόχθονες σε κάποιες ε, περιοχές. Εγώ είχα πάει σε μια περιοχή πολύ απομακρυσμένη όπου όλοι οι κάτοικοι είχαν ε, κινητά. Ε, θα πρέπει να περιστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέσω επικοδομητικής συνεργασίας και ε, πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή πραγματικά είναι ιδιαίτερως επίκαιρη. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι με ανησυχεί πάρα πολύ ένα ιδιαίτερως πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποφελθούν κάποιοι ξύπνοι θα πρέπει να έχουμε μια λογική προσέγγιση και να απλοποιήσουμε το σύστημα αυτό ή δυνατόν. Κάτι που βεβαίω δεν είναι πάντοτε εύκολο. Αλλά πραγματικά θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε πέντε λεπτά. Paul Murphy. Επόμενος είναι ο Πολ Μέρφυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια. Εάν διαβάσει κανείς τις τροπολογίες, ε, διαπιστώνει κανείς ότι πιάνουν σε διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις και υπάρχουν δύο ξεκάθαρες ε, γραμμές, ως και περισσότερες ε, διαφορές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συνένεση, είναι μάλλον απίθανη. Από τη δική μας άποψη, είναι, το θέμα είναι κατά πόσο θέλουμε σοβαρά να ασχοληθούμε με τη μείωση των ρήπων του διοξεδίου του άνθρακα, κατά πόσο θέλουμε να οδηγηθούμε σε κάποιες συνέπειες όσον αφορά τα συμβατικά βιοκαύσιμα και να πάρουμε σοβαρά αυτές τις οδηγίες ασχολούμενοι με αυτά τα ε, θέματα. Το ζήτημα δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. και τα σημεία κλειδί κατά την άποψή μου είναι καταρχήν η θέσπιση ενός κατοφλίου 5% ε, για τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Η Επιτροπή προτείνει ένα κατόφλι της τάξης του 3%. Δεύτερον, όσον αφορά αυτό τον παράγοντα iLook, ε, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί η οδηγία, θα τεθεί σε ισχύ, με την ε, ενίσχυση των κριτηρίων ε, βιωσιμότητας, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα δικαιώματα των αυτοχθόνων, την υφαπαγή γης, το δικαίωμα για τροφή κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεύτερον, η ενίσχυση του συστήματος επαλήθευσης της συμβατότητας, του ελέγχου συμβατότητας ε, και διασύνδεση με την εργασία που έχει γίνει στο παρελθόν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και τρίτον, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα σε σχέση ή ένα ερωτηματικό μάλλον σε ποιο βαθμό ορισμένα από αυτά τα προϊόντα τα οποία περιγράφονται ως ε, προωθημένα, προηγμένα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, πράγματι πληρούν αυτά τα κριτήρια. Και ορισμένοι ζητούν να αποσυρθούν ε, από τον ε, κατάλογο βάσει αυτού του παράγοντα πολλαπλασιαστή, γιατί νομίζω θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για τα ωφέλη αυτών των προηγμένων βιοκαυσίμων πριν προωθηθούν ειδικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ανοίγουμε τη σύντηση με τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Ο κύριος Λάγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν τότε θεσπίστηκε αυτή η ποσόστοση του 10% εγώ ήμουν ξεκάθαρα κατά. Γιατί διαπίστωσα ήδη ότι με τέτοιου είδου ποσοστώσει ε, μπορούν να γίνουν εσφαλμένε λάθο επενδύσει. Αλλά με επέκριναν με δρυμή τρόπο πάρα πολλοί οργανισμοί του προστασία του περιβάλλοντο, ε, λέγοντα όλο να υπονομεύσω την προστασία του περιβάλλοντο. Τώρα αντιστρέφεται η κατάσταση, τώρα με επικρίνουν γιατί θέλω να εγγυηθώ την ασφάλεια της ε, επένδυσης, των επενδύσεων στα υφιστάμενα καύσιμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να οργανωθεί έτσι η μετάβαση, ώστε οι επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει να μπορούν μακροπρόθεσμα να παραμείνουν σταθερές. Αλλιώς θα ε, χαθούν πολλές θέσεις απασχόλησης και δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβατώ με μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε μια βραδία μετάβαση προς τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Δεύτερον, ε, το θέμα των εισαγωγών ε, θα το ρυθμίσουμε όπως ε, το ζήτημα της παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν τα, οι ποσοστώσεις για τα βιοκαύσιμα να πληρούνται μέσω εισαγωγών ε, που, προϊόντων που έχουν παραχθεί κάτω από βέβαιες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε η ποσόστοση των καυσίμων να μην χρησιμεύει στην εισαγωγή βιοκαυσίμων από τρίτες χώρες που έχουν παραχθεί υπό αμφίβολε συνθήκε. Και αυτό ισχύει και για την υποστήριξη των εξαγών. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, η βιοεθανόλη, η οποία πάει από τη Βραζιλία στι Ηνωμένε Πολιτείε, στη συνέχεια ε, βάσει του προτιμησιακού καθεστώτος να εξαχθεί και πάλι από τις Πολιτείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένας φαύλος ε, κύκλος, τον οποίο δεν θα πρέπει να στηρίξουμε. Και ένα τρίτο σημείο ε, η σήμανση ε, χρησιμοποιημένων ε, χρησιμοποιημένου λαδιού για βιοκαύσιμα δεν στέκει. Για παράδειγμα στο Βέλγιο όπου υπάρχουν όλες αυτές οι τηγανιτές πατάτες τις οποίες θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Αν το γενικεύσουμε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επινοήσουμε μία βιομηχανία αξιοποίησης του χρησιμοποιημένου λαδιού και θα τονώσουμε τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. και πρέπει να ευχαριστήσει τον κύριο Λάγκε. Ναι, θα τον ευχαριστήσω με τη σειρά του. Θα προσπαθήσω να είμαι απλός. Όπως ξέρετε είμαι καλλιεργητής. Ε, και δεν ε, καταλαβαίνω ποιο είναι το σύστημα υπολογισμού. Όσον αφορά τη δεύτερη γενεά, ε, τα προηγμένα βιοκαύσιμα, συμφωνώ με σένα, Μπέρντ. Στο βαθμό που έχουμε ρευστά καύσιμα και το καίμε σαν ε, θερμαντικό έλεο δεν, ε, δεν έχει κανένα νόημα να παράγουμε ρευστά καύσιμα από βιομάζα. Γιατί η βιομάζα έχει το όταν χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς έχει την υψηλότερη τιμή. Και εδώ μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ε, θερμαντικό λάδι. Αλλιώς ε, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την, τον ενθουσιασμό που υπάρχει για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Ε, θα φτιάξουμε από άχυρο ρευστά καύσιμα. Εμείς χρειαζόμαστε το άχυρο για το, για, την ποιότητα του, για να ισχύσουμε την ποιότητα του εδάφους. Ε, υπάρχουν άλλα πεδία που θα είχε νόημα αυτή η χρήση. Και εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τους πράσινους, γιατί εδώ είναι κατά της ε, δημιουργίας ε, καυσίμων. Wenn Από αραβόστο Εάν ε, έχουμε τέσσερις ε, τόνους ε, αραβόσιτο και 1,7 έλαιο αραβοσίτου και έχουμε μια καλή στρατηγική στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε περιφερειακά με την ε, ελαιοκράμβη να έχουμε καλά αποτελέσματα. δεν μπορώ να καταλάβω τους πρασίνους. Η ελαιοκράμβη είναι ένας από τους καλύτερους ε, ε, καρπούς που έχουμε. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια εκτάρια καλλιέργειες ελαιοκράμβη στην Ευρώπη. με την ελαιοκράμβη δεν έχουμε καθόλου διάβρωση. Έχουμε πλήρη κάλυψη του εδάφους και προσπαθούμε να καταστρέψουμε αυτές τις καλλιέργειες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και ε, θεωρώ ότι οι επιστήμονες οι οποίοι βοηθούν σε τέτοιου είδους, υποβοηθούν τέτοιου είδους προσπάθειες δεν αξίζουν αυτό το χαρακτηρισμό. Πριν πάμε στην εισηγήτρια, ας ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Φάνστιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την πολύ καλή έκθεση που συνέταξε. Ε, ήταν επικοδομητική η συζήτηση το απόγευμα σήμερα και βλέπουμε ότι το θέμα αυτό έχει προσελκύσει και τη δική σας προσοχή και το κατανοούμε. Είναι σημαντικέ και οι εμπορικέ πτυχέ διεθνώ που σχετίζονται με το ντοσχέ αυτό και να μην το ξεχνάμε. Κατά πρώτον, να πούμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συμμεριζόμαστε απολύτω την άποψη που εκφράστηκε ότι οποιαδήποτε λύση και αν προκρίνουμε για να αντιμετωπίσουμε το iLook θα πρέπει να μπορεί να σταθεί στο διεθνές ε, επίπεδο, ιδίω στον ΠΟΕ. Αυτό το καθορίζουν και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ανάλυση και η μελέτη αντικτύπου είναι ένα από τα κριτήρια που εφαρμόσαμε. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το σέβεται επαρκώς αυτό και χρήσιμο θα ήταν να σχολιάσω εν συντομία τι ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως για τα κατόφλια, ε, τα ανώτατα όρια. Τι σημαίνουν τα ανώτατα όρια στην πράξη. Το πρώτο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για κατόφλι ανώτατο όριο, για το πόσα πρώτη γενιάς βιοκαύσιμα μπορούν να καταναλωθούν ή πόσα τέτοια καύσιμα μπορούν να παραχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Είναι ένα ανώτατο όριο για το πόσα βιοκαύσιμα πρώτη γενιάς θα μπορέσουμε μέσω των ευρωπαϊκών οδηγιών να προκαλέσουμε να παραχθούν, να χρησιμοποιηθούν ω μέρο τη ενεργειακή μα πολιτική. Αν είναι 5% το ανωτοτόριό μα, δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Α το ξεπεράσουν αν θέλουν. Και ω προ την παραγωγή και ω προ την κατανάλωση καυσίμων πρώτη γενιά. Ούτε σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν δικαίωμα να προβλέψουν κρατική ενίσχυση για βιοκαύσιμα πρώτη γενιά πέραν του 5%. Το μόνο που σημαίνει το 5% είναι ότι ως κράτος μέλος δεν μπορείς να καταμετρήσεις πάνω από 5% για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Τα επιπλέον βιοκάψιμα του στόχου του 10% θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να είναι προηγμένης μορφής, δεύτερης ή τρίτης γενιάς βιοκάψιμα. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο δεν έχει σκοπό η πρόβλεψη αυτή ούτε να εμποδίσει την εξέλιξη των βιοκαυσίμων, εφόσον επιθυμούν τα κράτη-μέλη να τα προωθήσουν. Απλώς θέλουμε να διαχειριστούμε τα κίνητρα που παράσχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, για το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί, το μοντέλο παραγωγής, γιατί τέθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά. Είμαστε σαφείς όταν εκφράσαμε το μοντέλο και το πόσο εύρος το θέλουμε να αυτό το μοντέλο όπως παρουσιάζεται από την πρόταση. Οι, οι τιμές του iLook και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αρκετά σταθερά ώστε να χρησιμοποιηθούν και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο αυτό για να αποφασίσουμε ποια βιοκαύσιμα είναι βιώσιμα ή όχι και ποια θα έπρεπε να παίρνουν κρατική επιχορήγηση ή ενίσχυση ή όχι. Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά σταθερό ώστε να περάσει μηνύματα και προς την αγορά μέσω της διαφάνειας και της υποβολής εκθέσεων που τα κράτη-μέλη θα οφείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτής για την ποιότητα των καυσίμων. Για τον λόγο αυτό νομίζω ότι ήδη αντιλαμβανόμαστε ότι αβεβαιότητες υπάρχουν βέβαια για το μοντέλο μας. Εν όμως τις οποίες δεν θα αντιμετωπίσουμε έτσι αυτομάτως. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή σας, κάποιες ε, δεν θα αποπειραθώ καν να τις σχολιάσω. Σε καμία περίπτωση όλες. Απλώς ε, ορισμένες να θίξω. Πρώτα απ' όλα πώς ε, καταμετρούμε την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αυτά που λέει η οδηγία δεν αφορούν μόνο τα βιοκαύσιμα, αλλά τις ανανεώσιμες πηγές και τα καύσιμα για μεταφορές. Λόγω χάρη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Αυτό θα καταμετράτε. Και μάλιστα πολλαπλώ Μας απασχολεί απλώ αν η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στα τρένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να καταμετρηθεί πολλαπλασιαστικά, διότι τότε θα καταστεί και ενό νοήματο ο στόχο του 10%. Ήδη σήμερα το έχουμε, αν τα μετρήσουμε έτσι. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια στα τρένα. Και ανανεώσιμε πηγέ για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Οπότε θα είχαμε πετύχει ήδη το στόχο μα και δεν είναι αυτή ακριβώ η πρόθεσή μα. Συμφωνούμε ένα πρόσθετο πολλαπλασιαστή για τι οδικέ μεταφορέ να χρησιμοποιηθεί εφόσον οι πηγέ είναι ανανεώσιμε. Αυτό θα παράσχει επιπλέον κίνητρα για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα λόγω χάρη, αλλά όχι ηλεκτρική ενέργεια για άλλα κοινωνιακά μέσα. Λίγα λόγια για κάποια άλλα από τα σημεία που εφήγησαν στη συζήτηση. Ε, χρήση και η ιδιοκτησία γης έχει υποβάλει έκθεση σχετικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση πρόοδου που δημοσίευσε στα τέλη Μαρτίου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι προς στιγμήν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η επιπλέον ζήτηση βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει αρνητικά ενδεχομένως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας γης ή την χρήση της γης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και να το ελέγχουμε. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω για την πολλαπλή καταμέτρηση. Αυτό το βρίσκουμε σημαντικό για να περάσει ένα σαφές μήνυμα και προς την αγορά. Ότι υπάρχουν δηλαδή βιοκαύσιμα στα οποία πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη αξία, υψηλότερη τιμή. Αυτά δηλαδή που παράγονται από προϊόντα που δεν απαιτούν ε, τη χρήση γης. Κατάλοιπα και απορρίμματα κυρίως αλλά και φύκια. Φύκια που δεν ε, επηρεάζουν τη χρήση της γης. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Να αποφύγουμε την ε, υπερβολική τη χρήση της γης για να παράγονται βιοκάψιμα. Αυτά είναι τα σημεία και εκεί ήταν οι βασικές μας μέρημνες ε, και θέλαμε να σχολιάσουμε εφόσον κάποιες τροπολογίες από αυτές που προτείνονται εγκριθούν. Ευχαριστούμε. Τελικές παρατηρήσεις από τον εισηγήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο, όσους συμφωνούν ε, λίγο λιγότερο ή πολύ λιγότερο. Ε, το θέμα είναι ότι έχουμε μείωση παραγωγής τροφίμων, έχουμε την ε, απερίμωση των δασών ε, σε τρίτες χώρες από τις οποίες αγοράζουμε κάψιμα, μείωση, ανάγκη μείωση των εκπομπών διοξιδίου. Εδώ όμως μιλάμε για το σύστημα. Το άλλο κλαίτε, είναι εύρωστο, είναι πολύ συμπαγές κτλ. Δεν λέμε ότι δεν είναι. Το θέμα είναι το μοντέλο. Είναι το μόνο μοντέλο Μήπως σε άλλα πανεπιστήμια υπάρχουν άλλα μοντέλα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως επέλεξε η Κομισιόν, θεωρεί ότι είναι κατάλληλο και το έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Για να μην συνεχιστεί αυτή η απερίμωση των δασών και για να μην χρησιμοποιούνται γέες που είναι ε, ουσιαστικά για την καλλιέργεια τροφίμων, για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Το δεύτερο θέμα είναι αν έχουμε αυτές τις πολλαπλές, τετραπλές αξίες για συγκεκριμένες ουσίες ή στοιχεία ή αν πλέον θα μιλάμε για ποσοστά. Αυτό που σας ανησυχεί αλλά και εμάς είναι αυτό που λέγεται ε, ότι πρέπει να γίνει μελέτη επιπτώσεων, ότι πρέπει να προασπιστούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει, παράγουν και μας λένε και οι ίδιες επιχειρήσεις ότι θα ήθελαν. Θα μου πει η Κομισιόν αν ε, απατώ. Ότι δεν έχουμε πλέον περάσει την παραγωγή των καυσίμων δεύτερη γενιά, αλλά αυτό θέλουμε να προωθήσουμε, την παραγωγή καυσίμων δεύτερη γενιά. Θα πρέπει να δώσουμε κάποια περιθώρια για τα καύσιμα πρώτη γενιά και για τα καύσιμα δεύτερη γενιά. Αυτό με τον ηλεκτρισμό ωραίο μα φάνηκε, αλλά για την Κομισιόν βλέπουμε να μην ισχύει το ίδιο με αυτού του πολλαπλού υπολογισμού κτλ. Είναι τεχνικό το ζήτημα, πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά πρέπει να μας ξεκαθαρίσει η Κομισιόν, γιατί πρέπει να δώσουμε στην αγορά ένα πάρα πολύ ξεκαθαρό μήνυμα. Δηλαδή ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τις γέες, δεν θέλουμε να καλλιεργούνται βιοκαύσιμα σε γέες που ουσιαστικά πρέπει να καλλιεργούνται για την παραγωγή τροφίμων και επίσης θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ δεν σας κατάλαβα πολύ καλά και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το σημείο γιατί είναι αρκετά πολύπλοκο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πράγματι επίμαχο, πράγματι αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας στην επόμενη τακτική συνεδρίαση που έχουμε τον Ιούνιο. Και περνάμε στο σημείο 25. παρουσίαση της έκθεσης αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στο Τρινιδάδ και τον Πάγκο για την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κάρι Φόρουμ Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία Οικονομικής Σχέσης με την περιοχή Κάρι Φόρουμ. David Μάρτιν, εισηγητής, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να θυμίσω στους συναδέλφους, παρακαλώ, παρακαλώ, να θυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτή η Επιτροπή ακριβώς επέμεινε να έχουμε την οικονομική εταιρική σχέση καρυφόρου με Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η μόνη αυτή τη στιγμή επίσημη τέτοια συμφωνία και θέλαμε να δούμε την εξέλιξή της. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ήταν στις Βρυξέλλες το 2011. τότε, τώρα μάλλον όπως είπατε, συναντηθήκαμε στην Τρινιντάρ και τον Μπάγκο. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη η συνάντηση από τους οικοδεσπότες μας και με, με υψηλό ποσοστό προσέλευσης από τους ε, ενδιαφερομένους και εταίρους. Υπήρχε μια μικρή αντιπροσωπεία έξι ευρωβουλευτών οι οποίοι όμως ήταν όλοι πολύ δραστήριοι κατά τη συνάντηση ε, και είχαμε και εξαιρετική στήριξη από το προσωπικό μας. Στην πρώτη σύνοδο ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διοργάνωση, τους κανόνες, το modus vivendi της Επιτροπής και θα σας ικανοποιήσει το γεγονός ότι πέραν της Συμβουλευτικής Επιτροπής όλες οι υπόλοιπες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κανονικά. Συμφωνήσαμε λοιπόν για την εσωτερική διοργάνωση ως προς το ποιος θα προεδρεύει, ε, στην κάθε επιτροπή σημαντικά ζητήματα και μετά περάσαμε στα σοβαρότερα ζητήματα. Η δεύτερη σύνοδος ξεκίνησε με παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή της Καριφόρουμ, η οποία ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Χαρήκαμε με τη δουλειά που έχει κάνει και δεν θα ήταν αδιακρισία να πούμε ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής είναι ε, φοβερά επαγγελματία και πολύ υπεύθυνο και έθιξε αρκετά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, τις δασμολογικές περικοπές και την ανησυχία του για το ποσοστό περικοπής τους. Τι γίνεται με τα παλαιά οχήματα και το χαρτί δεν λύσαμε κάποια από τα ζητήματα, διότι η άποψη ήταν ότι είναι πολύ σαφείς οι διατάξεις για τις θεσμολογικές αυτές περικοπές και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα, όσα είχαμε υποσχεθεί μέσω του Aid for Trade δεν επετέφθησαν. Η θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την διαφοροποίηση και τη μελλοντική βοήθεια μπορεί να επηρεάσει τη στήριξη προς τις χώρες της Καραϊβικής και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτιστικές, στην πολιτιστική παραγωγή και τις, τους σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Εκπαίδευση, αθλητισμός, εθνική κληρονομιά και ούτω καθεξής είναι τα ζητήματα που διέπονται από αυτά ε, τα μέτρα και μας ενδιαφέρουν και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε περισσότερο οικονομικά από όσα παράγονται εδώ και όχι μόνο σε αυτές τις χώρες. Το κοινοβούλιο, όπως είπα, είχε έντονη παρουσία στις συζητήσεις και θίξαμε και το θέμα των απαιτήσεων θεωρήσεων για τους πολίτες ε, της Καραϊβικής που έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν ήταν άμεσα συσχετιζόμενο με την Συμφωνία Οικονομικής εταιρική σχέση, αλλά απασχόλησε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στο παρελθόν. Είναι όμω και θέμα εμπορική που έχει εμπορική διάσταση, γιατί οι πολίτε που δεν μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν και την εμπορική δράση των χωρών αυτών. Στη δεύτερη σύνοδο είχαμε παρουσιάσει από τον τομέα των κατασκευαστικών υπηρεσιών, αρχιτεκτονική, εθίγησε μια σειρά από προβλήματα για τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από την οικονομική τέτοια σχέση και καταγράψαμε και κάποιον ενθουσιασμό και αισιοδοξία για το μέλλον τη ε, συμφωνία αυτή, εφόσον υλοποιηθεί πλήρω. Τέλο, Πρόεδρε, επισκεφθήκαμε το Πανεπιστήμιο του Τρινιντάτ και τον Πάγκο. Τονίσαμε τη σημασία της παιδείας για την όλη περιοχή με την ε, παροχή προσωπικού ε, εξειδικευμένου προσωπικού στην περιοχή αυτή και την έλευση φοιτητών από εκεί προ τα εδώ, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά σχολιάσαμε και τα θέματα τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πόρων, δηλαδή θα μπορούσαν να διοικητευτούν για να ανανεώσουν τι τουριστικέ υποδομέ. Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση των επικεφαλής ε, αντιπροσωπιών των Ευρωπαϊκών Πρεσβειών και εν είδη συμπεράσματος να πω Πρόεδρε ότι όλο το διήμερο πραγματικά ε, εκτελήχθηκε σε πολύ καλό κλίμα όλες μας οι συζητήσεις και σαφώς η οικονομική εταιρική σχέση δεν λειτουργεί ακόμη πλήρως ούτε δίνει όλα τα ωφέλη που αναμένει κανείς να αποδώσει. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Ε, θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να επαναλάβω τα όσα είπε ο Ντέιβιντ Μάρτιν ότι πραγματικά ήταν ένας εξαίρε... που ήταν ένας εξαίρετος πρόεδρος της αντιπροσωπείας και νομίζω το κλίμα μεταξύ ευρωβουλευτών ήταν υπέροχο. Και ήταν υπέροχη επίσης η οργάνωση εκ μέρους των, ε, ε, από τους οικοδεσπότες μας. Ε, αυτές είναι χώρες που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Μεταξύ αυτών ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών που δεν είναι ήδη σε όλες τις χώρες. Το CARICOM, το CARIFORUM, και λοιπά. Υπάρχουν ε, διάφορα είδη οργανισμών ε, σε κάποιες χώρες, άλλοι σε άλλους, αλλά ε, δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμοι και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία και πηγαίνουμε σε κάποια νησιά ή σε κάποια εδάφη τα οποία ανήκουν σε ευρωπαϊκές δυνάμεις και είναι τμήμα της Καραϊβικής. Τα, θέματα, τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν αναφέρθηκαν από τον David ε, Μάρτιν και νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη συνεργασία για την ανάπτυξη εκ μέρους της ε, Ευρώπης. Ε, εγώ βρίσκομαι σε μια Επιτροπή Συνεργασίας για την Ανάπτυξη και μας ανησυχεί, μας απασχολεί ιδιαίτερα στο θέμα των θεωρήσεων και εάν ε, καταργηθούν ε, οι θεωρήσεις αυτές ε, θα υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία, πολιτιστικές ανταλλαγές κλπ. νομίζω ότι ο Ντέβιτ Μάρτιν με κάλυψε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ευχαριστούμε. Κάποιο άλλο να σχολιάσει, η κυρία Ρινάλντι, ήσασταν και σήμερα μέλο τη αντιπροσωπεία. Ναι, να ευχαριστήσω και εγώ τον Ντέιβιντ για την αναδρομή και τα όσα μας είπε, είναι μια περιοχή που πραγματικά είναι συναρπαστική. Προνομιακές σχέσεις έχουν οι χώρες αυτές με πολλές περιοχές του κόσμου, με τις ΗΠΑ κατά πρώτον. Έπειτα είναι και τμήμα της νότιας, της λατινικής έστω Αμερικής και μετά και την Ευρώπη που την έχουν μακριά βέβαια, αλλά είναι ισχυρή πολιτιστική και ιστορική δεσμή με την Ευρώπη. Αυτό το συζητήσαμε, ψηφίσαμε το πρωί, συζητήσαμε και ψηφίσαμε και την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια για την μελλοντική συμφωνία με τι ΗΠΑ. Όμως η πολιτιστική συνεργασία, η πολιτιστική βιομηχανία και παραγωγή είναι κάτι που θα πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η οικονομική εταιρική σχέση καρυφόρμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ περήφανοι για την πολιτιστική του παραγωγή. Είναι θέμα ταυτότητα και είναι κάτι που έχουν και να πουλήσουν αλλά και κάτι να μάθουν από όλο αυτό και το καταλαβαίνουν. Και να τονίσω το ζήτημα των θεωρήσεων. Για αυτού είναι ύψη τη σημασία. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό. Σαφώ νομίζω ότι είμαστε στη, στο λάθο, στρατόπεδο, στο, στη λάθος πλευρά. Δεν υπάρχει θέμα μετανάστευση. Είναι άσχετο αυτό το θέμα. Και πρόκειται πραγματικά για διακριτική μεταχείριση των επιχειρηματιών του. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Ντέιβιντ, έχει να πει κάτι για να κλείσουμε. Ελ, μπορείς να μα πει τίποτε για τους βουλευτές της Καριφόρουμ παρακολουθούν την εκτέλεση τη συμφωνία. Πολύ καλή ερώτηση. Το κοινοβουλευτικό φόρουμ είναι διακοινοβουλευτικό. Κοινοβούλιο με κοινοβούλιο. Συμμετοχή όμω στη συνάντηση ήταν αθρώα, η προσέλευση δηλαδή, αλλά κάποιες φορές δεν είχαμε τους ίδιους τους υπουργού εμπορίου. Είχαμε υπευθύνους τους που γνωρίζαν πολύ καλά τα θέματα, αλλά όχι αναγκαστικά τους άμεσα αρμόδιους. Πάντως στο κοινοβουλευτικό φόρουμ βουλευτές είχαμε πολλούς. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών ασχολούνται με την οικονομική εταιρική σχέση Και παρόλο που οι βουλευτέ ήταν πολλοί, δεν μπορούσαμε να κρίνουμε κατά πόσον οι κυβερνήσει συνολικά ασχολούνται με το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε διακοινοβουλευτικέ ε, συναντήσει σε τέτοιου είδου συμφωνίε. Ε, έτσι μπορούμε να δούμε την επιτόπια εφαρμογή των συμφωνιών. Ωραία λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 26. Πρόεδρο των τριμερών διαπραγματεύσεων. Κανεί από του εισηγητέ δεν είναι εδώ. Όμως, εγώ έχω συμμετάσχει σε όλες τις τριμερείς διαπραγματεύσει. Οπότε να μιλήσω δύο λεπτά για το πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Για τον κανονισμό πλαίσιο, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και για τη μακροοικονομική βοήθεια είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Συμβούλιο και για τα δύο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την πρωτοβουλία για τον κανονισμό πλαίσιο. Παρόλα αυτά, οι δύο συνομοθέτες, Συμβούλιο και εμείς, συμφωνήσαμε να υπάρξει κάτι σαν εικονική συμφωνία και αποφασίσαμε να κάνουμε μια κοινή δήλωση για το θέμα της γεωργίας. Ε, ένα σπάρο, δυο τριγώνια δηλαδή. Και πουδού, που και γεωργία. Θα φροντίσουμε να συμπεριληφθεί συνολική συμφωνία μας με το Συμβούλιο ε, σε έναν κανονισμό. Γιατί είπαμε οι υπόλοιπε πρωτοβουλίε αποσύρθηκαν από την Επιτροπή. Ίσως και απόψε. Γιατί σε μισή ώρα πηγαίνω σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Και ελπίζουμε σε τελική συμφωνία, η οποία θα είναι ευπρόσδεκτη. Το θέμα αυτό δεν έβρισκε λύση. Για τα Omnibus 1 και 2, πολύ πρόοδος έχει επιτελεστεί χάρη στην Ιρλανδική Προεδρία, καλύφθηκαν πολλές από τις δικές μας απαιτήσει. Τώρα για το που μπουσένα. Μάλλον το 2. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Λάιχτφριντ, θα πρέπει να ανακοινώσει στο Συμβούλιο αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι. Πιθανότατα η ομάδα διαπραγματευτών θα πει ναι στην προσφατότερη πρόταση του Συμβουλίου. Ωστόσο, για το Omnibus 1, η κυρία Ρόβελ που είναι η συγγήτρια δεν είναι ακόμα σε θέση να πετύχει συμφωνία διότι η προσφορά του Συμβουλίου δεν μας ικανοποιεί. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος και δεν μας ικανοποιεί πλήρως σε κάθε περίπτωση παρόλο που έχουν κάνει πολλά, πολλές παραχωρήσεις. Και τα δύο θέματα είναι δεμένα μεταξύ τους, είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε το ένα από το άλλο, πρέπει να συμφωνήσουμε και στα δύο. Ακόμα δηλαδή και αν τα βρούμε στο Omnibus 2, θα πρέπει να περιμένουμε τη συμφωνία και για το Omnibus 1. Όμως η δική μου προσωπική εκτίμηση επειδή παρακολουθώ τις διαπραγματεύσεις από την αρχή-αρχή, είναι ότι η συμφωνία την πετύχουμε πριν το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας. Πραγματικά η Ιρλανδική Προεδρία έφερε ένα αεράκι φρεσκάδας στην διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή αυτό είναι ένα, αυτή είναι μια εύκολη νομοθεσία. Υπάρχουν καθόλου ερωτήματα. Μια, ε, ένα ελάσσον ερώτημα. Ε, θα ολοκληρωθεί το Omnibus 2 κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ας περιμένουμε να δούμε. Ε, πραγματικά έχω πιστοσύνη ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πρώτη φορά που η Κομισιόν αποσύρει μια πρωτοβουλία γιατί δεν της αρέσει ο τρόπος με τον οποίο οι νομοθέτες επιτυγχάνουν μια συμφωνία. Και είναι πρώτη φορά που οι νομοθέτες αποφάσισαν να πετύχουν μια συμφωνία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια κοινή διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει ένα κανονισμό. Δεν έχει άρθρα, δεν έχει τη μορφή ενός κανονισμού, αλλά υπάρχουν ήδη όλες οι δεσμεύσεις και σημαίνει ότι στο μέλλον όλες οι περιπτώσεις μακροοικονομικής συνδρομής θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με ένα σωστό τρόπο γιατί συμπεριλαμβάνονται στο κανονισμό πλαίσιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πετύχαμε μια πολύ θετική έκβαση για την Ένωση και για εκείνες τις χώρες που επίσης ε, επιθυμούν αυτή τη συνδρομή. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ιδιαίτερος ε, πρωτότυπο και εφόσον ε, δεν υπάρξουν ενστάσεις νομίζω ότι απόψε μπορούμε να έχουμε και μια επίσημη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το τέλος της συνεδρίασής μας. Όχι, έχουμε άλλο ένα θέμα της ε, δραστηριότητας εποπτικών ομάδων. Υπάρχει εδώ κάποιος υπεύθυνο. Ο Μπεντ για την Κολομβία και το Περού. Με δύο ο γιατί καμιά φορά γράφεται ε, το Κολομβίο όχι με δύο όμικρον αλλά με OU. Ίσως ε, αυτό επηρεάζεται από τη γερμανική παράδοση, όπου η Κολομβία είναι κολούμπιεν με U. Η εποπτική ομάδα συνεδρίασε και αποφασίσαμε ότι μετά τη σύναψη μιας εμπορικής ε, συμφωνίας θα παραμείνουμε παρόντες για να εποπτεύσουμε την εφαρμογή στην Κολομβία και στο Περού. Και κάθε δύο μήνες περίπου θα συνεδριάζουμε και καταρχήν ε, θα καλέσουμε τους δύο προσβευτές από την Κολομβία και το Περού, καθώς και την Κομισιόν, η οποία επίσης έχει αναλάβει την δέσμευση να συνοδεύσει όλη αυτή τη διαδικασία ε, και θέλουμε σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου το οποίο εγκρίναμε ένα χρόνο μετά τη θέση ισχύ της συμφωνίας αυτής να διοργανώσουμε ένα σεμινάριο με ε, τους εταίρους μας την Κολομβία και το Περού, ιδιαίτερα τους ε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να ελέγξουμε σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ. Νότιος Κάφκασος, υπάρχει κανείς όχι. Βιέτναμ. Βιετνάμ, όχι. Ινδία. Α, η Μαρία Μπαντία, Ινδία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη μέρα. Έχουμε κουραστεί, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Οι ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Ινδία είναι κάπως δύσκολες. Συνεδριάσαμε με την ομάδα αυτή, παρακολούθησα αρκετέ φορές. Αρκετά τακτικές ε, ομαλές ε, επαφές έχουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον πρέσβη έχουμε συναντηθεί άτυπα και στο Δελχή και στην Καλκούτα πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε μια επίσκεψη. Πριν σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Είναι λίγο ασαφή, είναι λίγο ρευστά Όλοι νομίζουν ότι δεν μπορούμε να περάσουμε ε, σε μια προθεσμία μετά τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, γιατί τον Απρίλιο του 2014 είναι εκλογέ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά ε, το ότι στην Ινδία γενικά η κυβέρνηση ε, δεν είναι πολύ σταθερή. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά από πολιτική πλευρά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κατάφερε να περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία, ιδίω ό,τι αφορά τι ασφάλειε και τι δημόσιε προμήθειε. Είναι σε κατάσταση, αν, για να μην πω παράλυση, αδυναμία να λαμβάνει αποφάσει η κυβέρνηση τη χώρα. Όπω γνωρίζετε, η κυβέρνηση έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα διαφθορά και είναι σε πολύ αδύναμη ε, κατάσταση θέση τις αρχές ή μέσα Ιουλίου θα μπορούσαν ενδεχομένως να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αν όμως υπήρχε ξεκάθαρο συμβιβασμός για συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να έχουν επιληθεί πριν την ε, οριστική υπογραφή. Αυτοί οι οποίοι απαιτούν την ε, νομοθεσία ενδεχομένως να μην μάλλον ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να υπάρξουν ε, κάποια νομοθετήματα, ίσως να μην υπάρχει χρόνος ακόμη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε την απόφαση. Το Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση, αλλά πρέπει να περιμένουμε το νέο Κοινοβούλιο. Και πριν υπογραφή θα πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανόν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν έχουν κλείσει ακόμα. Ένα από αυτά, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι η ε, αυτοκίνηση τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά και τα ενοπνευματώδη. ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά, μάλλον τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Και αν δεν υπάρχει μία πρόταση που θα μπορούσαν να αντιδεχθούν ε, και Ινδοί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Με όλα αυτά που σα είπα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει τελικά να περιμένουμε να εξαντλήσουμε όλε τι δυνατότητε ή δηλαδή τέλη ή μέσα Ιουλίου, όχι ίσως πιο πέρα, εκτός αν έχουμε κάποια πρόοδο. Μάλλον θα είναι δύσκολο. Στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο, τη δική μας και τη δική τους να υπογράψουμε τη συμφωνία, μάλλον κοινοβουλευτική περίοδο. Το monitoring group θα δούμε τώρα πώς προχωρά η διαπραγμάτευση, θα μπορούσε να προτείνει ένα ψήφισμα. Θα περιμένουμε όμως τα μέσα Ιουλίου για να δούμε τι ειδήσει έχουμε. Και μετά θα λάβουμε τελικά μια απόφαση, θα το συζητήσουμε γιατί είναι πραγματικά κρίμα. Πολλή δουλειά έχει γίνει ήδη και τώρα ε, δεν λέω να περιμένουμε το κοινοβούλιο, τη νέα κυβέρνηση και μετά και το δικό μας νέο κοινοβούλιο και μετά την νέα επιτροπή. Θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν σε μια τέτοια περίπτωση. Θα το δούμε να πούμε ότι ναι, έχει εκλογέ ε, στην Ινδία, αλλά και από τη δική μα την πλευρά υπάρχει ενδιαφέρον και γι' αυτό πρέπει και μετά να διαπραγματευτούμε. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. πρόεδρο. δεν ξέρω αν ε, συμφωνώ με την απεισοδοξία σου και αν τη συμμερίζομαι τέλο πάντων. Μερκοσούρη Χωσέφα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι ήταν μεγάλη μέρα σήμερα. Ε, έκαν, κάναμε λοιπόν ε, ένα ταξίδι με πρόεδρο τον Λουίς Γιάννφ ε, στην περιοχή αυτή και διάφοροι από τον Πυρίλο, η Άννα Μιράντα, η γομνική συγκήτρια. Ήταν ικανοποιητική η επίσκεψή μας σε ό,τι αφορά Ενδεχομένω νέε εξελίξεις. Πήγαμε στην Αργεντινή, πήγαμε στην Ουρουγουάη. Για να μιλήσω για την Ουρουγουάη πρώτα. Εκεί κάναμε πολλά και διάφορα. για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με την Ουρουγουάη. Υπήρξαν κάποιες ε, προτάσεις, κάποιες προσφορές από πλευράς ε, της Ουρουγουάης. Θεωρεί ο Ρουγά ότι χάνει εμπορική μερίδιο ε, στις εμπορικές δραστηριότητες. Ναι, για τον ε, Ουρουάη μιλάω. Χάνουν σε ανταγωνιστικότητα. Και οι πρέσβει το ε, και τα εμπορικά επιμελητήρια και των πολιτών, τα συνδικάτα και οι δημοσιογράφοι. Μιλήσαμε με όλους αυτούς. Ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον. Ο Πρόεδρος από πολιτικής και γεωστρατηγικής πλευράς μας χαρακτήρισε ως μία μονάδα εξισορρό... μία, μία μάλλον δύναμη εξισορρόπησης. Και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, να ε, έχει τη θέση της αναλογή. Επίσης μας κάνανε και ένα μάθημα φιλοσοφίας και το προσωπικό και μας είπε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μας είπαν ε, ουσιαστικά ε, με αυτά τα λόγια, ε, εάν δεν μας θέλετε υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Θεωρούν λοιπόν ότι η συμφωνία του Μερκοσούρ δεν είναι μόνο εμπορική συμφωνία, είναι μια συμφωνία αξιών, είναι μια ουσιαστική συμφωνία αφορά και τη δημοκρατική διαδικασία και είναι πολύ σημαντική. Τώρα, για την Αργεντινή, εκεί δεν ήταν τα πράγματα ακριβώ ίδια. Η κατάσταση στην Αργεντινή, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις εκεί. Είναι σε κατάσταση αυτοάμυνας, ε, εθνικιστική προσέγγιση, άρα ήταν διαφορετικό το πλαίσιο εκεί. Η κοινωνία των πολιτών βέβαια ενδιαφέρεται στη χώρα αυτή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ε, ευρωπαϊκή κρίση λόγω και της κρίσης στην Αργεντινή και τα συνδικάτα ε, ενδιαφέρονταν και υπήρχαν και πορείε τότε, λαλητήρια ήταν και πρωτομαγιά όταν ήμασταν εκεί. Τους ενδιαφέραν όλα αυτά τα θέματα που συζητούσαμε εκεί, ιδίως για την εμπορική συμφωνία. Όμως Ούτε η πρόεδρος της Αργεντινής ε, μας δέχτηκε. Αυτό είναι το ε, αρνητικό, αλλά ο Πρωθυπουργό ε, μας δέχτηκε, ο Καγκελάριος, όπως λέει, και μας έθεσε δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι με τη συμφωνία στον Ειρηνικό δεν έχουμε πρόοδο, το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κολομβία-Περού δηλαδή. Εκεί έχουμε κάποια ζητήματα ιδεολογικά, πολιτικά, τα οποία ε, παίζουν ρόλο και σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ είμαστε λίγο ε, σε μετέωρη κατάσταση. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη πάντως συμφωνία και οι Αργεντίνοι έθεσαν διάφορα ζητήματα, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τα δια γονιδιακά τα τραντζένιξ με τη ΣΥΠΑ, αν συμφωνήσουμε. Τους ανησυχούσε το θέμα, σε ενδιέφερε. Una valoración este fin de año Θα πρέπει επίσης να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου πώς θα προχωρήσουμε. Οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Πιέζονται και οι ίδιοι τους ενδιαφέρουν αυτές τις συμφωνίες οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν προχωρήσει και τώρα περιμένουν την κίνηση τη δική μας. Εμείς περιμένουμε η, η Βραζιλία η οποία θέλει να απελευθερώσει τον μπλοκ και κάνει μονομερείς συμφωνίες με την Αργεντινή όπως και η Ουρουάη με τη Βραζιλία. Ε, υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων διμερών συμβάσεων. Η Κίνα τώρα, ο Χέλμουτ Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα έχουμε μια συνάντηση της εποπτικής ομάδας, της ομάδας παρακολούθησης της 6 Ιουνίου, όπου θέλουμε να διαπραγματευτούμε ή να συζητήσουμε θέματα των συγκρούσεων των διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Κίνα, και Κίνας ως σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα καθώς και η Συμφωνία Επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Και με την ευκαιρία αυτή θα προσκληθούν όλα τα μέλη της Επιτροπής και επίσης οι συντονιστές να συμμετάσχουν. Νομίζω ότι πρόκειται να γίνει μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η επόμενη συνάντηση, εφόσον δεν υπάρχουν διάφορα, προσεχή συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Άντε. Άντε. Αμάν. Αμάν. Okay. I'll